Liebe, liebe Οι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας ε, καλωσορίσω. Äh, να σας καλωσορίσω σε αυτήν την ε, συνεδρία. Έχετε την ημερήσια διάταξη μπροστά σας. Υπάρχουν κάποιες επιθυμίες ή προτάσεις σε σχέση με την ημερήσια διάταξη για αλλαγές ίσως. Εφόσον δεν υπάρχουν εγκρίνεται. Υπό το σημείο 2 δεν έχω κάποια ειδική αναγγελία να κάνω ως πρόεδρος ή κάποια ανακοίνωση. Θέλω μόνο να σας πω για εκείνους που δεν το γνωρίζουν ακόμα ότι μια μικρή αντιπροσωπεία θα πάει στη Μεγάλη Βρετανία σήμερα το απόγευμα και αύριο θα έχουμε διαφορετικές συναντήσεις μεταξύ άλλων με μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και του Υπουργείου Οικονομικών της Bank of England και των κοινωνικών εταίρων. Περνάμε τώρα στο ουσιώδες, ουσιοδέστερο στοιχείο της σημερινής μας συνεδρίασης. Έχει αφιερωθεί αυτή σε μια ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους της ε, Γαλλικής Βουλής, του Γαλλικού Κοινοβουλίου. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να χαιρετήσω εδώ άμεσα εξ αριστερών, δηλαδή από εσάς δεξιά, τον κύριο Ανρί Εμμανουελή, είναι ο πρόεδρος chairman και σας διαβάζω τον τίτλο στα αγγλικά γιατί δεν τον έχω γερμανικά. Ο τίτλος είναι, δεν είναι εύκολο να μεταφραστεί, αλλά ευχαριστώ τους επαγγελματίες διερμηνείς μας που θα τα καταφέρουν. Ελπίζω να τα καταφέρουν κουτσάστραβα, Πρόεδρος της Επιτροπής Inquiry, Εξεταστικής Επιτροπής για το μηχανισμό, κερδοσκοπικό μηχανισμό σε σχέση με την μηχανισμούς και λειτουργία των οικονομιών. Δεν ξέρω αν έτσι είναι ε, σωστά ο τίτλος, αλλά αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, δίπλα του, από μένα αριστερά, για σας δεξιά, κάθεται δίπλα του Ζαν Φρανσουά Μανσέλ, ο εισηγητής αυτής της Επιτροπής της Γαλλικής Βουλής για την κερδοσκοπία. Να σας δώσω κάποιες επισημάνσεις για τη σταδιοδρομία και τα, την επαγγελματική του διαδρομή. Ο πρόεδρος είναι ο κύριος Εμμανουελή, πολιτικές επιστήμες σπούδασε στο Παρίσι και ήταν και στον κόσμο της οικονομίας που είχε δραστηριοποιηθεί στην εταιρεία, οικονομική εταιρεία Rothschild πριν από το... Ναι, βλέπετε, δεν είναι κάτι το αυτονόητο να εργάζεται κανείς στο Rothschild και το 1978 βουλευτής εξελέγει ως βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος και προσήθε στην Εθνοσυνέλευση, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και επανεξελέγει επανειλημμένα αρκετές φορές μετά από αυτή την ημερομηνία. Εν ήταν και υφυπουργός ήταν ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, ενδιάμεσα και τώρα είναι ακριβώς υπό την ιδιότητα του Προέδρου αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής εδώ. Ο γείτονα του Ζαν Φρανσουά Μανσέλ σπούδασε νομικά και στη συνέχεια πολιτικές επιστήμες και τέλος ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές ε, σπουδές του, στην École Nationale d'Administration, στην Εθνική Σχολή Διοίκησης ε, και έτσι πέρασε επίσης ε, στο Υπουργείο Υποδομών και Συντονισμού Σχεδιασμού και εκείνος εξελέγει ως βουλευτής επανειλημμένα κιόλας για την ΕΠΕΡ και μετά για το UMP Εν τω μεταξύ ήταν και δύο χρόνια ευρωβουλευτής εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μεταξύ 1984-1986 και ο πρώτος γραμματέας ήταν του κόμματος RPR 1995-1997 και τώρα είναι εισηγητής αυτή της εξεταστική επιτροπή. Έχουμε στόχο κατά το δεύτερο ήμιση των εργασιών της Επιτροπής μας να είμαστε σε επαφή με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είχαμε πάει στην Πράγα, Λισαβόνα, Μαδρίτη, τώρα θα πάμε στο Λονδίνο. Μετά έχουμε και μια αποστολή που θα κάνουμε στην Αθήνα. Μάλιστα. Και σήμερα για άλλη μια φορά συγκεκριμένες επαφές ε, είχαμε με το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας και φαίνεται ότι κατά το πρώτο ήμιση του Φεβρουαρίου πιθανώς ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια αποστολή και να έχουμε ε, εκεί και μια συνάντηση με τα μέλη της ε, Ομοσπονδιακής Βουλής. Να σας πω επίσης ότι οι απαντήσεις στις 7 συγκεκριμένες μας ερωτήσεις που είχαμε αποστείλει σε όλα τα 27 εθνικά κοινοβούλια αυτές τις 7 ερωτήσεις καλύτερα και πιο γοργά υποβάλλονται από ό,τι αναμέναμε ή ελπίζαμε κιόλας ή τολμούσαμε να ελπίζουμε. 10 ή 12 έχουμε απαντήσει. Κάποιε από αυτέ τι απαντήσει είναι πολύ εξειδικευμένε και σε βάθο και επακριβώ ασχολούνται με τα ερωτήματά μα. Και έτσι απορρέει από αυτό νομίζω μεγάλο input, πολλά στοιχεία πληροφόρηση που μπορούμε να αποκομίσουμε. Θα πρότεινα τώρα στη συνέχεια να ακολουθήσουμε την εξή διαδικασία. Καταρχήν να ακούσουμε τον κύριο Εμμανουελή που θα λάβει πρώτος τον λόγο. Μετά θα συνεχίσει με την παρέμβασή του ο κύριος εισηγητής Μανσέρ και οι δύο κύριοι σύντομα θα μας δώσουν μια ε, επισκόπηση των εργασιών τους και των συμπερασμάτων τους. Και μετά θα έχουμε στη συνέχεια ευκαιρία να συζητήσουμε και για αυτά τα επτά ερωτήματα τα οποία είχαμε αποστείλει, να συζητήσουμε για αυτά και φυσικά να δούμε και τα συμπεράσματα σε σχέση με τα όσα έχουμε ως στοιχεία στη διάθεσή μας. Θα έχουμε μετά τον γύρο ερωτήσεων, απαντήσεων και έτσι μετά με την περβάνσα θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Κύριε, έχετε τον λόγο. Είναι η σειρά σας κύριε Εμμανουελή να προσφωνήσετε τους συναδέλφους. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υποδοχή σας εδώ που μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε εργασίες της Επιτροπής σας. Πρέπει να είμαστε σύντομοι φαντάζομαι και το πιο ενδιαφέρον θα ήταν σίγουρα να καταφέρουμε να απαντήσουμε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής σας. Δημιουργήσαμε την εξαστική αυτή κοινοβουλευτική επιτροπή. Πρόκειται για μια δυνατότητα που έχει το κοινοβούλιο μας προκειμένου να μπορούμε να εξετάζουμε εις βάθος κάποια ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Στα πλαίσια της Εξεταστικής Επιτροπής μπορούμε να έχουμε διάφορους συμμετέχοντες, διάφορους ελεγκτές, οι οποίοι μάλιστα παίρνουν όρκο για τα όσα λένε. Δεν λειτουργούμε εμείς ακριβώς όπως τα αγγλοσαξονικά κοινοβούλια. Προσπαθούμε μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής να εξετάσουμε εις βάθος κάποια στοιχεία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι κερδοσκοπικοί μηχανισμοί, οι οικονομικοί κερδοσκοπικοί μηχανισμοί. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώθηκε και εμφανίστηκε η κρίση στην Ελλάδα και θελήσαμε εξ αρχής να γνωρίζουμε αν υπήρχαν κάποια κερδοσκοπικά κινήματα, κάποιες δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών δηλαδή οργανισμών που ενδεχομένως να είχαν επιταχύνει, να είχαν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της κρίσης αυτής. Πολύ γρήγορα στραφήκαμε προς πιο γενικές επισκοπήσεις όσον αφορά την κρίση αυτή καθ' αυτή, για την απαρχή της, Ακούσαμε πολλούς καθηγητές πανεπιστημίου για την κρίση αυτή, καθώς επίσης και πολλούς ε, επιχειρηματίες, τελέχη επιχειρήσεων. Ακούσαμε επίσης και εμπειρογνώμονες ε, των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Μελετήσαμε στη συνέχεια τους μηχανισμούς που ισχύουν σήμερα για την ρύθμιση, τη μη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών και πιστεύω ότι ε, το όλο εγχείρημα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Περίπου 40 ακροάσεις ε, κάναμε, 38 άτομα περίπου καλέσαμε. Άνθρωποι που ερχόντουσαν από ε, πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα, από διαφορετικές χώρες πολλές φορές. Προσκαλέσαμε ακόμα και άτομα που ερχόντουσαν εκτός της Γαλλίας, όπως σας είπα, και καταφέραμε λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Θα ήθελα να συνοψίσω κάπως τα συμπεράσματα αυτά και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι είμαστε κυρίως εδώ για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας. Ενδεχομένως ο κύριος Ζων Φωνσουά Μανσέλ να μιλήσει πιο διεξοδικά για τις προτάσεις που κάνουμε. Καταλήξαμε πάντως σε κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, μας αναστάτωσε πάρα πολύ, μας προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη το να ανακαλύψουμε τα πραγματικά ποσά για τα οποία μιλάμε. Θα έλεγα ότι ε, ανακαλύψαμε, και αυτό δεν το είχαμε δει τόσο πολύ στην επικυρότητα, ότι από το 2004 μέχρι σήμερα η ρευστότητα, η παγκόσμια στι χρηματοπιστικέ αγορέ παρουσίαζε μια αύξηση της τάξης του 15%, ενώ η οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίω ήταν μόνο 4%. Καταφέραμε κατά αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία μιας τεράστια κερδοσκοπικής φούσκας Μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε περίπου για 700.000 δισεκατομμύρια δολάρια, Αυτά είναι αν θέλετε τα OTC, τα, οι εξοχρηματιστριακές συναλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα παγκοσμίω. Μιλάμε για γιγαντιαία ουσιαστικά ποσά και καταλαβαίνετε βέβαια ότι από την άλλη καλούνται οι πολιτικοί θύνοντες να ρυθμίσουν αυτή την τεράστια αχαλήνωτη αγορά. Οι περισσότερες χρηματοπιστριακές συναλλαγές γινόντουσαν σε συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες τελικά συναλλαγές όσον αφορά τους τίτλους, τα χρεόγραφα, τις αξίες γινόντουσαν σε πλατφόρμες οι οποίες δεν υπόκεινται στο σύστημα του reporting σε πλατφόρμες για τις οποίες δηλαδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις διαφάνειας και υποβολής αναφορών. Επομένως ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει, να γνωρίζουμε ακριβά, ακριβώς ποια είναι τα ποσά τα οποία συναλλάσσονταν. Ουσιαστικά μας προκάλεσε, το παραλαμβάνω για άλλη μια φορά εντύπωση, το μέγεθος της κατάστασης. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε με έμεσο τρόπο να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε αντίθεση με τα όσα πιστεύουν ορισμένοι δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση αυτή. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εκκρεμότητα και αυτό γιατί οι χρηματοπιστωτικές αγορές ξέρετε ότι δημιουργούν ουσιαστικά κερδοσκοπικές φούσκες οι οποίες άλλοτε επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Στο παρελθόν είχαμε τις νέες τεχνολογίες περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων και το καθεξής. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά χρήματα, μεγάλη ρευστότητα η οποία κυκλοφορεί παγκοσμίω και επομένω δεν απομένει παρά να αναρωτηθούμε ποια θα είναι η επόμενη κερδοσκοπική φούσκα η οποία θα εμφανιστεί και ποια είναι η σχέση που μπορεί να υπάρχει με την πραγματική οικονομία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα, εξελιχθεί η κατάσταση, πώς θα καταφέρουμε να αποκαλύψουμε, αν θέλετε, όλα αυτά τα ποσά. Είδαμε επίσης τι έγινε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στο εθνικό επίπεδο. Κινούμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε ένα κοινό νόμισμα, ένα νέο νόμισμα το ευρώ. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμεί καταλήξαμε σε μια διαπίστωση που πιστεύω ότι είναι και κοινή διαπίστωση των ευρωπαϊκών αρχών. Η τελευταία οδηγία η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια οδηγία ιδιαίτερα δυσμενής θα έλεγα γιατί δημιούργησε πάρα πολλές παράλληλες πλατφόρμες συναλλαγής σε τίτλους και σε χρεόγραφα. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο ε, η αρχική πρόθεση της οδηγίας αυτής ήταν να, να, αποφύγει, να αποφύγει ουσιαστικά μια λανθασμένη συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών αγορών, να μην έχουμε δηλαδή τη δημιουργία κάποιων μπλοκ χρηματιστηριακών. Παρ' όλα αυτά ε, ξεπέρασε η οδηγία αυτή της αρχικές της προθέσεις και δημιούργησε τις διμενείς επιπτώσεις τις οποίες αναφέρθηκα. Και βλέπουμε ότι ε, πολλές φορές υπάρχει κάποια απόκληση ανάμεσα σε αυτά τα οποία μας είπαν οι προσκεκλημένοι μας. Υπάρχει το high frequency trading, για παράδειγμα, το οποίο εμείς θέλουμε να καταργηθεί. Υπήρχαν κάποιοι προσκεκλημένοι μας οι οποίοι μας είπαν ότι δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, δεν είναι τόσο σοβαρό. Και υπήρχε ένας άλλος προσκεκλημένος μας ο οποίος μας είπε ότι μα αυτό ακριβώς αντιστοιχεί περίπου στο ίμιση των ε, ποσών που ε, συναλλάσσονται στα χρηματιστήρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Καταλήξαμε πάντως εμείς σε κάποιες ε, προτάσεις, 20 περίπου. 34 συγκεκριμένα, για τις οποίες θα μας μιλήσει ο συνάδελφός μου, ο Ζωφρονσουά Μανσέλ, ο οποίος θα σας παρουσιάσει λοιπόν. Και στη συνέχεια βέβαια στη διαθεσή σας για ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ που μας προσκαλέσατε και μας υποδέχεστε εδώ. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ εγώ ιδιαίτερος, διότι μου θυμήσατε μια διετία ευτυχίας που πέρασα στο Ευρωκοινοβούλιο μεταξύ του 1984 και του 1986. Σχεδόν ε, μου στήχησε να επιστρέψω στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, διότι εδώ πραγματικά πέρασα μια διετία που με γέννησε ενθουσιασμό. Ε, όχι μόνο γιατί υπήρξα βουλευτής, αλλά γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων εδώ. Τώρα, ας έρθουμε στις βασικές μας μέρημνες. Πώς, όπως είπε ο κύριος Μανουέλη πριν από λίγο, η εξεταστική αυτή επιτροπή δημιουργήθηκε βάσει πρόταση ψηφίσματος ε, που υπέβαλε το ε, σοσιαλιστικό μας κόμμα σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο του νέου μα κανονισμού ο πρόεδρος ε, της ομάδας που κατέθεσε την πρόταση ψηφίσματος ε, όρισε έναν εισηγητή, εισηγητή της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή την ε, πλειοψηφία εκπροσωπώ εγώ. Εργαστήκαμε λοιπόν από κοινού ε, σε τέτοιες συνθήκες που καταλήξαμε το σύνολο των κομμάτων που συνέμεριχαμε σε αυτήν την τριανταμελή επιτροπή να βρεθούμε στο πέρα των εργασιών να εγκρίνουμε ομόφωνα την έκθεση τη Εξεταστική Επιτροπή. Την έκθεση αυτή λογικά την έχετε στη διάθεσή σα, ιδίω ω προ τι προτάσει τη. Ε, το θέμα αυτό δεν ε, άφησε αδιάφορο το Ευρωκοινοβούλιο στο πλαίσιο των ζητημάτων που και σας αποσχολούν. Ο κύριος Εμμανουέλη μίλησε για τις ακροάσεις που οργανώσαμε, τις προσωπικότητες που υποδεχτήκαμε και προσκαλέσαμε, ιδίως ε, δίγνωστά μέλη της Επιτροπής σας, την Περβάνς Μπερές που βρίσκεται μπροστά μου ακριβώς και τον κύριο Γκοζές. Και οι δύο ήρθαν να μας δώσουν τη μαρτυρία τους στην ε, Επιτροπή την Εξεταστική μας και ολοκληρώσαμε και με την ακροάση ενός Ευρωπαίου Επιτρόπου, του κυρίου Μπαρνιέ. Έτσι λοιπόν ε, θεωρούμε ότι όσο το δυνατόν περισσότερο Ήμασταν ε, συντονισμένοι και συμβαδίσαμε με τις ε, ανησυχίες και τις μέρημνες που και εσείς έχετε εδώ. Τώρα για τις γραμμές που δώσατε εσείς ε, στην εξέταση του θέματος και ο κύριος Εμμανουελή το ίδιο, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και να πιστέψω την προσοχή σας σε ορισμένες από τις προτάσεις μας. Έχουμε κάνει 34 προτάσεις και δεν θέλω να σας ε, καταπονήσω με την ανάγνωση 34 προτάσεων, όμως θέλω να σταθώ σε ορισμένες από αυτές που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε συζήτηση να σκεφτούμε και να μελετήσουμε το όλο θέμα. Όλος ιδιαίτερος ε, με ενδιαφέρουν οι ε, ευρωπαϊκοί διάστασεις διάστασης ανησυχία σας. Έχετε λοιπόν τις προτάσεις μπροστά σας. Σας ε, λέω λοιπόν να κοιτάξουμε μαζί την τέταρτη πρόταση που μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Εκεί προτείνουμε καλύτερη πολυμερή επαγρύπνηση από τα ευρωπαϊκούς φορείς για τις πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί από κοινού με τα κράτη-μέλη και ιδίως για, για το διαφορετικό ταμείο ε, και την επιρροή που μπορεί να έχει σε ορισμένα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί από κάποιους, μπορεί να προκαλέσει συζήτηση, αλλά είναι σημαντικό να το δούμε. Στην πρόταση 5 έχουμε ένα σημαντικό μέτρο, γιατί εδώ δεν μας ενδιαφέρει απλώς να στρέψουμε το βλέμμα μας στον συστημικό κίνδυνο του οικονομικού συστήματος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνδυνος τέτοιο μπορεί να υπάρχει στο εσωτερικό της Ένωσης ούτως ή άλλως. Όμω πρέπει να εργαστούμε σε πλήρη ε, συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Διότι όταν κοιτάζουμε πώς ξεκίνησε η κρίση, πώς πυροδοτήθηκε, ε, καθίσταται προφανές ότι οι γύροι ελέγχων που κάνουμε ε, θα πρέπει να βασίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Εάν τέτοιες διαδικασίες ελέγχου, όπως τις οργανώνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, δεν αντιστοιχούν σε αμερικανικούς ελέγχους... Ε, θα έχουμε μια δυσκολία και μια πλέον δυσκολία αν δεν υπάρχει ανταλλαγή των στοιχείων που συγκεντρώνουν οι ΜΕΝ και οι ΔΕ. Φανταστείτε το ενδεχόμενο μια μελλοντική κρίση αύριο σε διεθνέ επίπεδο θα υπάρχουν ε, συνέπειε. Και να θυμίσω εδώ και του στόχου του G20. Θα πρέπει να υπάρχει ικανότητα, δυνατότητα μάλλον διεθνώ αμοιβαίω να επικοινωνήσουμε και να προλάβουμε του ενδεχόμενου κινδύνου ε, μια επανάληψη τη κρίση. Τρίτο σημείο το οποίο βρίσκω και αυτό πολύ σημαντικό και εδώ νομίζω στην καρδιά των ερευνών των ε, Ευρωβουλευτών σε ό,τι αφορά δηλαδή την διαφάνεια στις αγορές. Πρόεδρε, πρόσεξα προηγουμένως ότι το ερωτηματολόγιο που υπενηχθήκατε, αλλά που ε, δεν έλαβε εγκαίρω η δική μα Εξεταστική Επιτροπή, διότι ολοκλήρωσε το έργο του στο Δεκέμβριο του 2010. Υπάρχει θέμα για του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μα, στην πρόσφατη παρουσίασή του, για, όταν μάλιστα έδωσε τις ευχές του στο διπλωματικό σώμα στο Παρίσι, ε, είπε ότι το θέμα αυτό τον ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Είναι λοιπόν ε, ωραία ιδέα για τον φόρο, αλλά όπως είπε προηγουμένως και ο κ. Εμμανουέλη, έχουμε ένα σημαντικό όγκο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μας είπαν στην Επιτροπή μας ότι το 50% των διεθνών χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών ξεφεύγουν της ε, επαγρύπνησης των επίσημων φορέων δεν είναι γνωστέ. Πώ λοιπόν να επιβάλλουμε φόρου μόνον σε όσου είναι μέσα το παιχνίδι, είναι νόμιμοι, διότι όσοι μένουν εκτό και είναι αδιαφανεί θα ξεφεύγουν. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα οικονομική αρχικά διαφάνεια και ανάγκη να θέσουμε από τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών το σύνολο των οικονομικών φορέων και το σύνολο των συναλλαγών. Αυτό είναι επιτακτική ανάγκη και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρέμβουμε. Εδώ έχουμε πράγματι καταμετρήσει τις αρνητικές συνέπειες των αρχικά καλών προθέσεων που είχε η οδηγία για τις αγορές και τα οικονομικά μέσα. Η οδηγία αυτή φαίνεται ότι δημιούργησε έναν, κάποιες δυσκολίες μη επιθυμητές και αρκετέ ω προ την διαφάνεια. Έχουμε τι ε, προτάσει 7 και 8 για το θέμα αυτό που βρίσκουμε ιδιαίτερα σημαντικό. Και θέλουμε και τη δική σας άποψη σχετικά, διότι θέλουμε να δούμε πώς βλέπετε την εξέλιξη της ενδεχόμενης ε, επαναθεώρησης αυτής της οδηγίας. Κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί και πριν το τέλος του καλοκαιριού 2011. Και για να παραμείνω σύντομος, Δύο ακόμη παρατηρήσεις μόνον. Η πρώτη αφορά ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα προσφυλές στη Γαλλία, το πρόβλημα της ρύθμισης των αγορών στο σύνολο των αγορών πρώτων υλών, ιδίω για τις γεωργικές τιμές. Εδώ έχουμε την πρόταση παριθμών 9, η οποία προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη ρύθμιση των αγορών. Για το σημείο αυτό έχουμε διαπιστώσει ότι βρισκόμαστε σε καθυστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ ακριβώς. Θα έπρεπε λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο ταχύτερα. Και τέλος, και εδώ σας θέτω εγώ ένα ερώτημα, ένα ερώτημα που μας, μας απασχόλησε ιδιαίτερος, το, η πλαισίωση των εναλλακτικών ε, συναλλαγών και κοντιλιών. Εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσπαθούμε να εγκρίνουμε τέτοια εναλλακτικά ταμεία και κονδύλια. Όμω αυτό μα απασχολεί ιδιαίτερα στην εξεταστική μα επιτροπή. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο που θα προβλέψουμε θα είναι εθνικό και επικυρωμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπω ε, κινδυνεύει τελικά να μην, εκπροσωπ... να μην περιλαμβάνει όλε τι απαραίτητε εγγύσει ώστε τα εναλλακτικά αυτά ταμεία να συμμορφώνονται με τι ευρωπαϊκέ ε, επιθυμίε. Να λοιπόν, ε, εν είδη εισαγωγής κάποιες ερωτήσεις και να, οι συστάσεις που κάναμε σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη της χρήσης. Διότι ξέρουμε πλέον τι πρέπει να αποφύγουμε σε σχέση με το παρελθόν, αλλά είμαστε και ρεαλιστές και πιστεύουμε ότι τα ίδια πράγματα μπορεί να ξανασυμβούν. Θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε πέραν των ευρωπαϊκών και ατλαντικών συνόρων και να σκεφτούμε ότι αύριο μπορεί να ξεκινήσει μια κρίση από την Ασία. Ποια θα είναι η δική μας δυνατότητα ώστε να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά κύριε για αυτές τις ακριβέστατες τοποθετήσεις από πλευρά σας. Για το έργο σας και τα αποτελέσματα θα ήθελα θερμά να σας ε, συγχαρώ. Και είδα και το εκτενές αυτό χοντρό βιβλίο ως αποτέλεσμα των ε, εργασιών σας. Ευχαριστούμε πολύ και για αυτές τις ε, προτάσεις που εξειδικεύσατε. Θα πρότεινα ως εξής να συνεχίσουμε. Καταρχήν, σε αυτές τις τοποθετήσεις που μόλις μας κάνατε, συγκεκριμένα να επισέλθουμε και να διατυπωθούν ερωτήσεις. Και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Στη συνέχεια μετά, σύντομα, να συνοψίσουμε ποια είναι τα δικά μας σύντομα συμπεράσματα εν συντομία και σε σχέση με αυτές τις επτά ερωτήσεις που είχαμε διατυπώσει και τις απαντήσεις που πήραμε. Καταρχήν θα έλεγα είναι καλύτερο να αρχίσουμε με την εισηγήτρια, την Περβόνς. Παρακαλώ και τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτής της ανταλλαγής απόψεων, η οποία θα μας επιτρέψει και εμείς να πάρουμε το λόγο και να εμπνευστούμε για τη συνέχιση των εργασιών μας στις προτάσεις που κάνετε. βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που έχουμε καλύψει και εμείς την δική μας την έκθεση. Η δική μας έκθεση βέβαια καλύπτει ένα πιο ευρύ πεδίο, δεν ασχολείται μόνο με την κερδοσκοπία. Όσον αφορά πάντως πιο συγκεκριμένα την κερδοσκοπία, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία καλύπτουμε και εμείς στην έκθεσή μας, ιδίως όσον αφορά την επαναδιπραγμάτευση της οδηγίας ε, MIF. MIF. Καταλαβαίνετε ότι η αρμόδια επιτροπή στο Κοινοβούλιο θα είναι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Πάντω η οδηγία αυτή συνέβαλε πολύ στην λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και οδήγησε ουσιαστικά και αυτή συνέβαλε στην κρίση. Επίση ε, είναι σημαντικό να δούμε ποια ρύθμιση μπορεί να υπάρχει για τι αγορέ αυτέ, οι οποίε παρουσίασαν πολύ μεγάλα κέρδη κατά τη διάρκεια τη κρίση. Αναφερθήκατε επίσης στο ζήτημα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ξέρετε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς ε, ψηφίσαμε για το ζήτημα αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια τέτοια φορολογία χωρίς να περιμένουμε να συμβεί κάτι τέτοιο σε παγκόσμιο επίπεδο. Ερχόμαστε σε επαφή με διάφορους συνομιλητές για το ζήτημα αυτό και συναντούμε και διάφορα εμπόδια. Είπατε κι εσείς ότι περισσότερες συναλλαγές οι χρηματοπιστωτικές παραμένουν αρκετά θολές, αδιαφανείς. Ιδίως στα πλαίσια αυτού του dark pool στο οποίο αναφερθήκατε. Μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα όντως, αλλά αν είχαμε τελικά μια φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, θα υποχρεώναμε τον νομοθέτη να τροποποιήσει, να διορθώσει την κατάσταση αυτή και να μην υπάρχουν πλέον αδιαφανείς συναλλαγές. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είχαμε και μια καλύτερη και μεγαλύτερη διαχείριση της ε, ανάληψης κινδύνου, η οποία γίνεται μέσω αυτών των συναλλαγών. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταφέρναμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε συστημικό κίνδυνο. Και αν εφαρμόσουμε μάλιστα και τα συμπεράσματα του G20, δεν θα είχαμε πλέον αγορές ή συναλλαγές οι οποίες δεν θα ήταν διαφανείς. Αναφερθήκατε επίσης σε κάποια πράγματα σχετικά με την πρότασή σας την υπαριθμό 18. αναφέρεστε εδώ πέρα στις ε, κεντρικές τράπεζες, στην ευθύνη που φέρουν. Και είπατε όμως ότι ανάλογες προτάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και, σε, και για άλλους οργανισμούς. Αναφερθήκατε στο ρόλο των οίκων αξιολόγησης, πώς επηρεάζουν τα πράγματα με την βαθμολόγηση την οποία δίνουν. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μια διπλή δυσκολία. Καταρχάς, οι οίκοι αξιολόγησης πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες αρχές όπως αυτές που έχουμε από την Επιτροπή της Βασιλείας. Ξέρετε ότι οι αξιολόγησεις έχουν αναλάβει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και η Επιτροπή της Βασιλείας τελικά με τον ένα την άλλο τρόπο ενσωμάτωσε κάπως την ιδέα αυτή, δηλαδή ότι οι διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν μόνο υπόψη τους τα όσα λένε οι ότι μετράει ουσιαστικά μόνο η βαθμολογία τους. Ενώ εμείς ε, στην ε, Βασιλεία 2, δηλαδή στην ε, πρώτη οδηγία CRD, όσον αφορά την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είχαμε πει ότι θα πρέπει να κοινοποιούνται όλες αυτές οι βαθμολογήσεις και μάλιστα να αξιολογούνται σε σχέση με άλλες μελέτες ή αναλύσεις που έχουν γίνει. Η ρυθμιστική λοιπόν αρχή, η Επιτροπή της Βασιλείας, παραχώρησε αυτή τη στιγμή μια αρμοδιότητά της στους οίκους αξιολόγησης και από την άλλη βέβαια έχουμε και τον τρόπο με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές αγορές χρησιμοποιούν στη συνέχεια την αξιολόγηση αυτή, τη βαθμολόγηση. Ο Προεδρός μας, υπό άλλη του αρμοδιότητα, ήταν εισηγητής για το ζήτημα αυτό και εγώ με τη σειρά μου υπέβαλα κάποιες τροπολογίες ακριβώς επειδή ήθελε η στάση μας να είναι λίγο πιο συνεπής και ελπίζω ότι ε, ο εισηγητής, ο πρόεδρός μας θα τις λάβει υπόψη του. Υπόψη του. Πάντως και το ζήτημα αυτό των οίκων αξιολόγηση είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ και στην πρότασή σας 26 ε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αναφέρεστε εδώ πέρα στις συμφωνίες της Βασιλείας και λέτε ότι θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να γίνουν ε, διεθνείς συνθήκες προκειμένου να βρισκόμαστε σε ισότιμο επίπεδο με τους ε, Αμερικανούς εταίρους μας. Αν ε, το Γαλλικό Κοινοβούλιο μπορούσε πραγματικά να υποστηρίξει την πρόταση αυτή, αυτό θα ήταν ε, ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεν έχω να κάνω άλλες παρατηρήσεις. Μία ερώτηση μόνο θα ήθελα να θέσω ποια είναι η άποψή σα για τη δική μα τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά δηλαδή τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Εν μέρη απαντήσατε. Πάντω με την άδειά σα κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω ότι η δική μα η έκθεση η οποία ουσιαστικά βγαίνει λίγο έξω από την στενή αρμοδιότητα τη δική σα Εξεταστική επιτροπή που ασχολείται μόνο με την κερδοσκοπία. Θα ήθελα να αφαιρθώ λοιπόν στη δική μας την έκθεση σε σχέση με το G20. Η Γαλλία ετοιμάζεται να λάβει την προεδρία του G20 και θα ήθελα ως προς αυτό να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, στο πλαίσιο αυτό τίθεται και το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Είχε απασχολήσει ιδιαίτερα την επικαιρότητα στο παρελθόν το ζήτημα αυτό. Ήταν από τα πρώτα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει ατονίσει λίγο προσοχή ως προς τους φορολογικού παραδείσους. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναλάβουμε δράση προκειμένου ουσιαστικά να βάλουμε κατά των περιοχών εκείνων που συμβάλλουν πάρα πολύ στην κερδοσκοπία, όπου η κερδοσκοπία υλοποιείται. Τι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει το G20 για το ζήτημα αυτό, για να το προωθήσει λίγο περισσότερο. Δεύτερον, θα αναφερθώ σε μία δέσμευση που αναλάβαμε στην συνεδρίαση του Pittsburgh, νομίζω, όπου είπαμε ότι κάθε αγορά, κάθε προϊόν θα πρέπει να υπάγεται σε ένα καθεστώς εποπτείας Και πάλι τώρα ως προς αυτό αναφερθήκατε κι εσείς πριν από λίγο όταν μιλήσατε για τις αδιαφανείς αυτές συναλλαγές, για τα dark pool, τις παράλληλες αυτές συναλλαγές. Και ως προς αυτό λοιπόν υπάρχει μια σημαντική δυσκολία. Είδαμε πώς η αγορά των CDS εκτοξεύθηκε Όταν ήρθα εγώ στη δική σας επιτροπή, σας είπα ότι ε, όλοι λένε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο ορισμός για την κερδοσκοπία και αυτό επιτρέπει σε κάποιους να λένε ότι δεν υπήρξε κερδοσκοπία στην Ελλάδα. Βλέπουμε όμως ότι οι κερδοσκόποι αστικά υποφελούνται ενός συστήματος αγοράς που έχει ήδη αρχίσει να ισχύει. Ενδεχομένως ε, να επωφελήθηκαν λοιπόν κάποιοι από μια ανισορροπία που υπήρχε στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας. Υπήρχε μια λογική της αγοράς η οποία μπορεί να οδήγησε σε υποβάθμιση της βαθμολόγησης της Ελλάδος και στη συνέχεια όμως είδαμε ότι υπήρξαν πολλοί χρηματοπιστωτικοί παράγοντες οι οποίοι επωφελήθησαν της κατάστασης αυτής ακριβώς για να προχωρήσουν σε κερδοσκοπικές συναλλαγές. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να επενθυμίσουμε τις δεσμεύσεις του G20 προ αυτό και μια τρίτη παρατήρηση Πώ μπορούμε να ακολουθήσουμε έναν ενιαίο δρόμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεσή μα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωζώνη θα πρέπει να εκφράζονται με μία κοινή ενιαία φωνή σε διεθνέ επίπεδο. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό αν πραγματικά θέλουμε να μπορούμε να μιλήσουμε με πυγμή όσον αφορά την πολιτική ε, τη της, της ισοτιμίας. Και δεν ενδιαφέρομαι εδώ πέρα μόνο στις σχέσεις δολαρίου και γιουάν. Το λέω για να είμαστε πάντα σε θέση ισχύω οποιαδήποτε και να είναι η κατάσταση του ευρώ. Πρέπει να μπορούμε να μιλάμε με μία ενιαία φωνή αν πραγματικά θέλουμε να μας ακούνε. Συγγνώμη που μακρηγόρησε, Θέλω να μιλήσω και για τις δικές σας παρατηρήσεις και για τη δική μας την έκθεση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εδώ θα, πω, θα κάνω λίγα σχόλια γιατί φύγεται ε, τον βασικό προβληματισμό για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι η ομοσπονδιακή διάσταση ή αν θα ακολουθήσουμε μια και μόνη οδό. Αυτό είναι πολιτική επιλογή, δεν είναι οικονομικό θέμα. Εάν υπάρχει μια και μόνη οδός, θα πρέπει να λειτουργεί με δημοκρατικά κριτήρια. Διότι αν η μόνη οδός που θα ακολουθήσουμε δεν βασίζεται σε πολιτική ισότητα, υπάρχει πρόβλημα. Είναι όμως πολιτικός ο προβληματισμό. Δεν είναι νομισματικός. Και ξέρουμε πολύ καλά από και από άλλα παραδείγματα ότι το ενίο νόμισμα για να είναι ισχυρό χρειάζεται πολιτική στήριξη πολλών. Εδώ έχουμε κληρονομήσει μια ιστορία την οποία δεν μπορούμε να επινοήσουμε εκ νέου. Ε, Βεβαίω έχουμε συμβάλει και εμεί στην δημιουργία τη, αλλά δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Και προσωπικό μου σχόλιο είναι, όχι τη Επιτροπή ολόκληρη, ότι καλό θα είναι να προσέξουμε να μην ακολουθήσουμε μια και μόνη οδό εάν δεν ακολουθήσουμε ισχυρού δημοκρατικού μηχανισμού που να εκπροσωπούν τι κοινέ γνώμε. Διότι εάν υπάρχει απόκληση μεταξύ κοινή γνώμη και μία οδού, θα υπάρχει πολιτική κρίση. Χωρί λοιπόν τι κατάλληλε δημοκρατικέ δομέ, τέτοια ε, μοναδική οδό δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου άποψη και δεν μπορώ να δεσμεύσω βεβαίω ούτε την άποψη των συναδέλφων, ούτε τη υπόλοιπη Επιτροπή. Τώρα, είναι θέμα κοινή λογικής. Κάναμε τόση δουλειά, τόσες με προσπάθειες και διερωτώμεθα μετά γιατί η κοινή γνώμη στην Γαλλία, στη Γερμανία. Φαίνεται να μην πιστεύει πλέον στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό ιδεώδε. Υπάρχει ένα, ένα ουσιαστικό πρόβλημα εδώ στην Ευρώπη, ένα πρόβλημα ουσία Είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό δημοκρατικό. Και το λέω εδώ αυτό ενώπιον των βουλευτών, γιατί ακριβώς το Ευρωκοινοβούλιο είναι ο τόπο όπου δημοκρατικώς εκπροσωπούνται οι πολίτε. Τώρα, Εάν μπορώ να κάνω πάλι μια προσωπική παρατήρηση και το λέω για τον ε, συνάδελφο Κλίντ, εδώ ήμουν ε, εκπρόσωπο του κόμματό μου για, τα, ε, για τι ευρωπαϊκέ υποθέσει και όταν έθεσε το θέμα αυτό μου ότι είναι υπερβολικά νωρίς. Τη στιγμή που ψηφίστηκε, ψηφιζόταν το Σύνταγμα, ήμουν κατά του συντάγματο, διότι για αυτήν τη φεντεραλιστική προσέγγιση του δημοσπονδιακού τύπου ε, μου έλεγαν πολύ αργά. Τη μια είναι πολύ νωρί, την άλλη είναι πολύ αργά. Τι να πω, ε, έχω γίνει πια ευέξατος για το θέμα αυτό. Τώρα, για τι υπόλοιπε παρατηρήσεις, για τον αφορό των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το συζητήσαμε, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Εγώ έχω πει ότι είμαι υπέρ. Όμω θα πρέπει όλα να βρίσκονται υπορρύθμιση, διότι εάν Μόνο όσοι πηγαίνουν στους επίσημους φορείς και υποβάλλουν τις εκθέσεις που απαιτούνται, ε, δεν κάνουμε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας φορός που να υποχρεώνουν όλους να δηλώνονται. Αλλά τίποτα δεν είναι βέβαιο βάσει των ευρωπαϊκών ηθών. Ε, δηλαδή κάποιοι μπορεί να πληρώνουν, κάποιοι όχι. ή για κάποιες υποθέσεις κάποιοι να πληρώνουν, κάποιοι άλλοι όχι, αλλά κατά επιλογή. Δεν, ε, τίποτα δεν είναι απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει αυτόματα. Όμως, για την ιστορία αυτή του φόρου, αυτού του περιβόητου, θέλω κάποιος να μου εξηγήσει τι συμβαίνει. Δηλαδή, από πολιτικής άποψης, δεν θα έπρεπε καν να το σκέφτομαι, αλλά διαρωτώ με, θέλουμε να φορολογείται η ρύθμιση ή η χρηματοδότηση της συνεργασίας των πολυεθνικών. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι χρήσιμο θα είναι γιατί είμαι ειδικό εισηγητής ε, στη Βουλή μας ε, για τις ε, εξαγωγικές πιστώσεις για τις χώρες, τις αναπτυσσόμενες, τις αφρικανικές. Το θέμα είναι αυτός λοιπόν ο φόρος ότι θα χρησιμεύσει. Τι θα ρυθμίζει. Υπάρχουν πολυάριθμες υποθέσεις όπου υπάρχουν ολόκληρη ολόκληρα ντοσχέ, η κωδική των φόρων είναι φάκελοι τόσο παχής δηλαδή να είστε σίγουροι αν προβλεφθεί τέτοιος φόρος δεν θα εμποδίσει τη φοροδιαφυγή ούτε γίνεται να βρούμε ως εκθαύματος καινούργια έσοδα πηγές εσόδων για μένα ε, τέτοιος φόρος σημαίνει τέρμα στην κερδοσκοπία και ρύθμιση στο σύστημα στο επίπεδο των διεθνών αγορών. Ε, ψηφίστηκα πρόεδρος της Επιτροπής ε, Οικονομικών, μάλλον ε, ψήφισα τον φόρο Τόμπιν τον, ψήφισαν δύο χώρε, η Γαλλία, ο Καναδά και κανεί άλλο. αυτό όταν ήμουν πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων το 2001. Λοιπόν, με αυτή τη συμβολική ψηφοφορία ανέβηκε λίγο το ποσοστό. Όμως, ακόμη και αν είναι πολύ χειρέ οι δηλώσει του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εγώ πολύ θα ήθελα να μου εξηγήσουν τι ακριβώς ε, προσδοκούν όλοι αυτοί που τα προτείνουν αυτά. Ε, και κάτι άλλο που δεν ακούστηκε αρκετά είναι το θέμα του reporting των εκθέσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να τα αποσπάσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τίποτε ε, χωρί τα πρώτα βήματα να είναι σωστά. Πρώτο είναι να γνωρίζουμε και για, ακούστηκε για τους φορολογικούς παραδείσους. Εγώ ανήκω σε τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα ε, στη Γαλλία που ε, μεταξύ Γερουσίας και Βουλής φαίνεται να είναι στην ίδια θέση που είναι η, ε, η Άνω και κάτω Βουλή της Γερμανίας. Λοιπόν, κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιες προτάσεις που μπορούσαν να περάσουν, κάτι φαινόταν ότι πάει να γίνει, όμως η κυβέρνηση δίστασε. Τώρα δεν θέλω εδώ να κατηγορήσω τη μια ή την άλλη κυβέρνηση για τη δράση της. Είναι πια αργά, αλλά δεν προχωρήσαμε γρήγορα, διότι οι συμφωνίες που ψηφίστηκαν για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και λένε απλώ ότι δεσμευόμαστε ε, να δίνουμε πληροφορίες για να βγούμε από τον μαύρο κατάλογο, εντάξει. Αλλά μετά πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί αυτό στην πράξη. Αυτό δεν ξέρουμε. Υπάρχουν χώρες όπως η Ελβετία που μας λέει συστηματικά όταν ζητούμε πληροφορίες υπάρχει προθεσμία. Μάλλον υπάρχει αδίκημα. Ναι, φοροδιαφυγή. Ε, για αυτούς δεν είναι αδίκημα η φοροδιαφυγή. Εντάξει, φαίνεται να υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά πρέπει κανείς να θυμώσει και να υψώσει τους τόνους. Ε, δεν είναι αυτό τώρα στάση. Επίσης εδώ δεν υπάρχει κανεί να μα ακούσει, έτσι. Δεν μας ακούει κανείς. Διότι οι Ευρωπαίοι υποτίθεται δεν αντρέχουν σε πρακτικές ε, φορολογικών παραδείσων. Εγώ δεν μπορώ να κατονομάσω κανέναν, αλλά υπάρχουν κάποιοι. Κάποιοι είναι πιο γνωστοί, κάποιοι λιγότερο, να δούμε τα αποτελέσματα. Να θυμόμαστε και την Εβάδα και το Ντέλαουερ. Εντάξει, αλλά δεν θα πω πώς λέγονται. Και ειδικά ναι, ένα τέτοιο παράδεισο σα είναι ιδιαίτερα προσφυλή, αγαπητέ Πρόεδρε, έτσι. Από την πλευρά του πατέρα σας. Όχι μάλλον από την πλευρά του πατέρα σας, αλλά της μητέρας σας. Τέλος πάντων, αυτά μπορεί ο καθένας να τα ερμηνεύσει όπως θέλει. Πρέπει να υπάρχει φορολογική σύγκληση και να έχουμε λάβει όλα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αλλά αν ακολουθήσουμε αυτήν την μία και μοναδική οδό, χωρίς να έχουμε πρακτικές συγκλίνουσες, χωρίς ανεπανομοιότητες, αλλά κυρίως τα φορολογικά και κυρίως την φορολόγηση των αποταμιεύσεων, και των συναλλαγών, ε, τα όρια θα είναι πολλά και πολύ περιοριστικά. Δεν χρειάζεται τώρα να σας πω πράγματα που ήδη τα ξέρετε παλού. Πολύ σύντομα για την φορολόγηση των συναλλαγών. Σημερίζομαι την ε, άποψη του κ. Εμμανουηλή. Είπαμε πολλά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής δεν θα άλλαζαν τα αποτελέσματα ως προς τον αγώνα κατά της κερδοσκοπίας. Δηλαδή, εάν οι κερδοσκόποι κερδίσουν από το κόστος των συναλλαγών τους, ανεβάσουν το κόστος των συναλλαγών τους, θα βγάλουν έτσι τη διαφορά για να πληρώνουν το φόρο. Άρα δεν θα είναι εισόδημα αναγκαστικά για μας. Πρέπει να αναζητήσουμε μια ευκαιρία να, να δημιουργήσουμε μια πραγματική πηγή νέων εσόδων. Για να είναι και επικοδομητικό αυτό το νέο μέτρο. Τώρα για τους φορολογικούς παραδείσους, εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξο από τον ε, Αρνή, ε, από τον Αρή για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι από το προηγούμενο G20 και ίσως και από παλιότερα, από το 2008, έχουμε επιτελέσει κάποια πρόοδο. Βεβαίως, όχι με το ρυθμό που αρχικά θυμούσαμε, αλλά σαφώς υπάρχουν κάποια βήματα πρόοδου. Στην έκθεσή μας, νομίζω στην υπαριθμό 3 πρόταση, ε, επενισόμαστε την εξέλιξη αυτή λέγοντας ότι είναι απολύτως αναγκαίο το G20 να ε, κάνει μια σφαιρική επισκόπηση των εξελίξεων των πολιτικών κατά των φρονικών παραδείσων. Και να μπορέσουμε βήμα προς βήμα να τα παρακολουθήσουμε αυτά, να έχουμε Τακτικέ συναντήσει για να βλέπουμε τι βήματα πρόοδο επιτελούνται. Σίγουρα δεν προχωρούμε με αρκετή ταχύτητα. Σίγουρα υπάρχουν ακόμη θύλακε φορολογικών παραδείσων. Σίγουρα εκεί ε, ευνοούνται οι κερδοσκόποι και η κάλυψη των εσόδων τους. Όμως ε, για να είμαστε βέβαιοι ότι θα προχωρήσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στον τομέα αυτό. Εδώ υπάρχουν τρεις ε, πολύ συγκεκριμένε προτάσεις και αυστηρές συστάσεις για τους ε, οργανισμούς πιστοληπτικής, εξελίξης πιστοληπτικής ικανότητας. Εδώ θα ανεβεί, ανέβει το θερμόμετρο, διότι κάποιες φορές θα θεωρήσουν κάποιοι ότι οι ενδείξεις που δίνουμε ε, δεν είναι ευχάριστες. Κάποιος καθηγητής οικονομολογίας Λοιπόν, πρόσφατα ε, που τον, ε, τον, τον οποίο συναντήσαμε μας είπε ότι δεν πέφτει από τον ουρανό η κερδοσκοπία. Οι οικονομικές περιστάσεις επιτρέπουν να ξεκινήσει να δημιουργείται μια τέτοια ροπή προς την ε, κερδοσκοπία. Και όλα τα παραδείγματα που έχουμε δει τώρα δείχνουν ότι η κερδοσκοπία γεννάται από καταστάσεις οικονομικές πολύ συγκεκριμένες που την προκαλούν εμέσως ή άμεσα. Επίσης, για τους οργανισμούς αξιολόγησης επιστολητικής ικανότητας που έχουν ε, τεράστιο ρόλο σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδίως για τους καινούριους, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να καλούνται να σεβαστούν έναν κώδικα δεοντολογίας πολύ πιο αυστηρό από αυτό που σήμερα ισχύει. Και από την άλλη θα πρέπει να ξέρουν ότι περιμένουμε από αυτές να αντιμετωπίζουν τα κράτη, τα εθνικά κράτη, διαφορετικά και μάλιστα αρκετά διαφορετικά από τους ε, ιδιώτες φορείς, τι ιδιωτικές εταιρείε. Αυτό αναφέρεται και στις τάσεις που κάνουμε, διότι θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να τα ανακατεύουμε όλα. Δηλαδή δεν είναι και τόσο αυτονόητο να εξισώνουμε ένα κράτος με έναν ιδιωτικό φορέα, μια ιδιωτική εταιρεία στο επίπεδο των χρηματοδοτικών συναλλαγών. Ε, ιδού ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις που θέλω να κάνω βάσει της παρέμβαση τη κυρία Μπερέ. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερω που συνεισέφερε ε, στην ενημέρωση τη Εκτελεστική μα Επιτροπή. Ε, Πρόεδρο, τώρα θα λάβουν τον λόγο αμέσω δύο συνάδελφοι, ο ένα μετά τον άλλον. Έτσι, δύο-δύο θα παρεμβαίνουμε. Τόμα Μαν μετά Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δύο συνάδελφοι στη μητρική τους γλώσσα τα εξέθεσαν και έχουμε και ένα πίνακα των προτάσεων στα γαλλικά. Κάπως γνωρίζω τα γαλλικά και θα σας το επιβεβαιώσει η Περβάνς που είναι πρόεδρο ε, μια ε, κοινοβουλευτική μα επιτροπή, Εγώ είμαι αντιπρόεδρο, μιλάμε καμιά φορά γαλλικά οι δυο μα. Κάποια σημεία ήταν σαφή, εντάξει. Είχαμε ακριβώ το θέμα με τον φόρο, το τέλο επί των συναλλαγών, χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Έχετε δίκιο κύριε Μανουελή, είναι διαφορετικά πράγματα, διαφορετικέ υποθέσει που θα τα ξαναδούμε όταν πρόκειται για τον ορισμό τέλους φόρου κτλ. Όμως η σκέψη, η βασική σκέψη είναι ίδια μέσω της γαλλικής πλευράς από το Σαρκοζή έχει επιβεβαιωθεί αυτό τελεσίδικα. Πρέπει να εργαστούμε από αυτής της πρότασης. Ερώτησή μου, αν οι Αμερικανοί δεν είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν, η πρότασή σας είναι να ξεκινήσουν οι Ευρωπαίοι να εργάζονται και να δώσουν συνέχεια ή όχι. Δεύτερη ερώτηση, ποιες υπηρεσίες. Ήταν σημαντικό θέμα για την ε, Επιτροπή για την εξέταση της κρίσης που είχαμε και υπάρχουν προτάσεις σε σχέση με τη Γερμανία να δούμε να δημιουργηθούν ευρωπαϊκοί οίκοι αξιολόγηση. Υπάρχουν και οι πρώτοι που έχουν αδειοδοτηθεί, πιστοποιηθεί. Η προπόθεση είναι πιστοποίηση για τον ευρωπαϊκό χώρο, τον χώρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επαρκεί για εσά. Τρίτη ερώτηση. Είπατε κύριε Μανουελή ότι το νόμισμα πρέπει πολιτικά να υποστηρίζεται. Απόλυτα σύμφωνο. Ένα από τα θεμέλια είναι ότι δεν θα διαπιστώνεται ένα σύμφωνο σταθερότητα μόνο, αλλά και θα τηρείται στη συνέχεια. Είναι πρόθυμη να δώσει μάχη για αυτό το σύμφωνο σταθερότητα που θα υλοποιηθεί η Γαλλία. Και όχι μόνο να υπάρχει, παρότι υπήρξαν παραβιάσεις στο παρελθόν ε, αυτού του συμφώνου και δεν έγινε τίποτα. Είσαστε υπέρ του να υπάρξει μια ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση ή επαρκεί για σας να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία μόνο. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Η Γερμανία και η Γαλλία το είδαν συχνά αυτό και έχουν συναντηθεί πολλές φορές και τώρα βρίσκονται πάλι δίπλα-δίπλα και προσπαθούν να, είναι ηγετι... να έχουν ένα ηγετικό ρόλο η Γαλλία και η Γερμανία. Εσείς πώς το βλέπετε. Ανήκετε σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα. Είναι εδώ θέμα, ας το πω έτσι, συμ... συνεργασίας μεταξύ δύο διαφορετικών στρατοπέδων ή απλά κάποιος πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία και κάποιοι πρέπει να ακολουθήσουν. Κάνατε μια ανάλυση για την κερδοσκοπία διαβάζω με μεγάλη ικανοποίηση το, το βιβλίο του Ζερόμ Κερβιέλ που ήταν υπεύθυνο ε, για μια μεγάλη κρίση που ξέσπασε στη Γαλλία για μια μεγάλη τράπεζα, ο Ζερόμ Κερβιέλ. Έχει κάποιε δικαιολογίε που αναφέρει. Λέει ότι έκανε πολλά ο ίδιο, αλλά οι προϊστάμενοι του δεν έλεγξαν τα πράγματα σε σχέση με το ποιοι κέρδιζαν ποια χρήματα και δεν παρακολύθηκαν οι εξελίξει. Και υπάρχουν και άλλα βιβλία για αυτή την κατάσταση. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η κατάσταση. Γίνεται κάτι στι μεγάλε τράπεζε σε εσά στη Γαλλία. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει μέρημνα ώστε οι trader, οι όσοι εργάζονται στο χρηματιστήριο να έχουν κάποια όρια, να έχουν κάποιου περιορισμού ή όχι. Να έχουμε όχι μόνο ε, θέσει από insiders, από ε, εσωτερικά εργαζόμενους εκεί, αλλά να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Τώρα στη συνέχεια θα ε, έχουμε άλλη μετά θα ακολουθήσει ο κύριος Όλε Σμιτ. Πολλές είναι οι ερωτήσεις για τον κύριο Κερβιέλ. Η άποψή μου είναι ανήκω στην αντιπολίτευση στη Γαλλία και κατά τη διάρκεια της α, πολιτικής μου ζωής ενστερνίστηκα διάφορες τοποθετήσεις ιδιαίτερα σκληρές θα έλεγα εναντίον του τραπεζικού τομέα ακριβώς επειδή ενδεχομένω τον γνωρίζω καλύτερα από τους άλλους επειδή έχω κινηθεί μέσα σε αυτόν ή τον γνωρίζω καλύτερα από άλλους. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι οι γαλλικές τράπεζες είναι από τις πιο ελεγχόμενες, ενδεχομένω οι πιο ελεγχόμενες στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει μια πολύ παλιά παράδοση στην ε, Γαλλία ήδη από το 1945 ότι είναι το κράτος το πλέον αρμόδιο όσον αφορά τις πιστώσεις που μπορούν να δοθούν, το ποσό δηλαδή το οποίο μπορεί να δοθεί με τη μορφή δανείων, το κράτος είναι που δίνει την πρώτη έγκριση και συνέχεια τα δάνεια αυτά περνάνε από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Ο κύριος Κερβιέλ διαχειρίστηκε 5 δισεκατομμύρια στα πλαίσια μίας συγκεκριμένη τράπεζας δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ εδώ πέρα τις γαλλικές ε, τράπεζες γιατί τις επικρίνω σχεδόν κάθε εβδομάδα στη χώρα μου. Επομένω δεν πρόκειται να αλλάξω εδώ πέρα τοποθέτηση μόνο και μόνο επειδή βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Πιστεύω πάντως ότι στα πλαίσια της κρίσης που, γνωρίσαμε οι γαλλικές τράπεζες δεν επηρεάστηκαν τόσο όσο, οι άλλες και αν κατάφεραν να αντισταθούν περισσότερο ίσως αυτό να οφείλεται και στο ότι δέχονται πολύ περισσότερο έλεγχο. Τώρα όσον αφορά τη συμφωνία Μέρκελ-Σαρκοζή δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε εδώ πέρα για μια πολιτική συμφωνία. Νομίζω ότι ο Μιτεράν και ο Κόλ συνονούνταν καλύτερα από ότι ο Σαρκοζή με τη Μέρκελ. Γνωρίσαμε και άλλες περιπτώσεις Ζισκάρ, Στάνερ, Σμιτ και ούτω καθεξής πολλές φορές ενδεχομένως ε, είναι και προσωπική υπόθεση ακόμα και η ίδια η συγκυρία. Ενδεχομένως τώρα η συγκυρία να βαραίνει πολύ περισσότερο από ότι οι προσωπικές συμπάθειες. Μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας λοιπόν πιστεύω ότι ε, το γνωρίζουμε και εμείς ότι μερικές φορές εκνευρίζουμε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες Όλο και περισσότερο ακούγεται ότι το γαλλογερμανικό αυτό ζεύγος κινεί την Ευρώπη. Είναι ένα ζεύγος όμως και αυτό η, ζωή αν θέλετε ενώ ζεύγους δεν είναι πάντα ανθόσπαρτη. Πολλές φορές γνωρίζουν προβλήματα και έτσι και εμείς. Το πρόβλημα λοιπόν της οικονομική αυτής διακυβέρνησης δεν είναι το αν θα πρέπει να λαμβάνει χώρα ή όχι, είναι ότι πρέπει να λάβει χώρα και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δημοκρατική συνένεση. Δεν θα πρέπει να φαίνεται ότι είναι απλώς ένα τεχνοκρατικό μέσο το οποίο αντικαθιστά την πολιτική βούληση ή ότι γίνεται το αντίστροφο. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Τώρα, το αν θα υπάρχει μία σύγκληση των μέσων ε, διαχείρισης όταν έχουμε ένα κοινό νόμισμα, νομίζω ότι αυτό εξυπακούεται. Διαφορετικά είναι σαν να μην γνωρίζουμε τι θα πει κοινό νόμισμα. Τώρα, το σύμφωνο σταθερότητας. Πάντα είχα τις αφιβολίες μου ως προς αυτό, γιατί ε, αυτό το οποίο σκεφτόμουν πάντα είναι ότι αν εμφανιστούν προβλήματα, κανείς δεν θα το σεβαστεί και ακριβώς αυτό έγινε στην πράξη οι δημοκρατικές κυβερνήσεις είτε ανήκουν στη δεξιά είτε ανήκουν στα αριστερά, ανεξαρτήτως πολιτικός φάσματος, λένε ότι ε, θα επιβάλλω δυσάρεστα μέτρα για την κοινή γνώμη μόνο και μόνο για να τηρήσω το σύμφωνο σταθερότητας. Μα αυτό δεν συμβαίνει ποτέ στην πραγματικότητα. Μόνο σε απολυταρχικά ολοκληρωτικά καθεστώτα μπορεί να να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα δημοκρατικά καθεστώτα δεν λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, επομένω όταν θεσπίζουμε κανόνες, οι κανόνε θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τηρούνται. Γιατί, γιατί αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένα ποσοστά όπως 60% ή 70% όσον αφορά το χρέος. Ε, η Ιαπωνία, ο Λίβανος βρίσκονται σε εντελώ διαφορετικά ποσοστά, επομένως ίσως είναι αυθαίρετο να θέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια τέτοια όρια. Οι κανόνες λοιπόν αυτοί, όταν τους θεσπίσουμε, δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ απόλυτοι και αυστηροί, γιατί στην περίπτωση αυτή δεν θα τηρούνται. Και αυτό ακριβώς έγινε. Αυτό έγινε στη Γαλλία, για παράδειγμα. Αυτό έγινε και στη Γερμανία κάποια στιγμή και αυτό θα μπορούσε να συμβεί και χτυπώ ξύλο να μην συμβεί, θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες χώρες. Γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή μια συζήτηση στη Γαλλία. Δεν συμφωνούμε στα πάντα με τον συναδελφό μου Μανσέλ. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για το αν θα πρέπει να αλλάξει το σύνταγμά μα, για το αν θα πρέπει να κινηθούμε περισσότερο προ το γερμανικό μοντέλο. Εγώ πιστεύω πω όχι, γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να ισχύσει ένα τέτοιο σύστημα. Δεν μπορούμε να προκαταβάλουμε την πραγματικότητα δέκα χρόνια νωρίτερα, θεσπίζοντα κανόνε. Σαφώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια οικονομική διακυβέρνηση. Θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένε κανόνες και να μην έχουμε και ψευδεστήσεις όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας. Θα δείτε ότι αν τυχόν μπούμε και εμείς σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση, δεν είναι απαραίτητα σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να τηρήσουμε πλήρως το σύμφωνο σταθερότητας. Ίσως είναι από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα θετήσουμε. Ίσως τα πράγματα είναι και πιο πολύπλοκα τελικά από ό,τι φαίνονται. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση το τελευταίο μέρος. Έρχομαι από μια μικρή χώρα εκτός Ευρωζώνης. Είμαι ένας από αυτούς που με ζήλο θέλουν η χώρα μου να ενταχθεί στην Ευρωζώνη. Πρέπει όμως να πω ότι οι τελευταίες σας παρατηρήσεις εδώ δεν είναι πιστικές ε, για τους πολίτες στη χώρα μας. Όταν είχαμε ένα δημοψήφισμα, αυτός ήταν, αυτό ήταν ακριβώς εκείνο το οποίο αναφερόταν. Οι, μικρές, οι μεγάλες χώρες δεν θα ακολουθήσουν τις αρχές του Συμφώνου Σταθερότητας ε, και θα δημιουργηθεί μια χαοτική κατάσταση. Διαρωτώ με λοιπόν, αν εσείς στην έκθεσή σας έχετε εξετάσει όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είσαστε πεπειραμένοι πολιτικοί, στην προηγούμενη φάση πριν ενταχθείτε στο ευρώ, οικοδομώντας το ευρώ είσαστε μέρος ή ξε, αυτών που ξεκίνησαν και τώρα είσαστε μέρος της κρίσης της ίδιας. Θεωρείτε ότι η Γαλλία και ίσως εσείς οι ίδιοι ίσως κιόλας έχετε κάποιες ευθύνες για να λογοδοτήσετε για όλα αυτά τα οποία τεκταίνονται και συνέβησαν. Δεν είναι μόνο για την αποτυχία της, των αγορών, είναι και η αποτυχία των πολιτικών ανδρών αλλά και πολιτικών που ακολουθήθηκαν από αυτούς τους πολιτικούς. Όταν πριν από δύο εβδομάδες στην Πορτογαλία ομολόγησαν ότι είχαν κάνει ολιστήματα και είχαν προβεί ολιστήματα και σφάλματα και στην Ισπανία μία ημέρα μετά ακριβώς είπαν όχι, όχι δεν κάναμε κανένα λάθος. Τα σφάλματα έγιναν από ε, όσον αφορά το συμβούλιο, συμβούλια για την ε, κρίση ε, subprime. Γιατί τα λέω αυτά. Δεν προσπαθώ με κανένα τρόπο να σας προσβάλλω ή να είμαι επιθετικός. Αντίθετα, πιστεύω ότι αν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά η Ευρώπη μακροπρόθεσμα με 27 κράτη-μέλη και 27 κράτη-μέλη στην ίδια την Ευρωζώνη κιόλα, διότι αυτό είναι θεμελιώδου σημασία να συμμετέχουν όλοι, πρέπει να μάθουμε να ακολουθούμε και να εφαρμόζουμε του κανόνε, να του σεβόμαστε. Αν δεν είμαστε πρόθυμοι να σεβόμαστε του κανόνε και του θεωρούμε ηλίθιου για άλλου να του ακολουθούν ή υπερβολικά δίσκαμπτου, ε τότε πώ θα μπορέσει κανεί να προσπαθήσει να ε, είναι σεβαστοί αυτοί οι κανόνες. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σας επ' αυτού. Άλλη μου ερώτηση τώρα. Κατάλαβα καλά όταν άκουσα ότι είπατε ότι θέλετε οι υψηλή συχνότητα χρηματηριακές συναλλαγές να καταργηθούν. Το είπατε αυτό, αλλά οι προϊστάμενοι λέει οι ανώτεροι δεν άκουσαν τέτοιες ε, προτάσεις και έτσι συνεχίστηκε η κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για το short selling και αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και τη Γαλλία και τη Γερμανία και ασχολούμαστε με αυτό το θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θέλουν να απαγορευτεί το short selling. Εσείς τι λέτε, είναι καλό το short selling για τις αγορές. Ίσως ακόμα και οι υψηλή συχνότητα συναλλαγές είναι καλές για τις αγορές. Τι λέτε. Ίσως σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες εγώ θα σας έλεγα αυτές οι τοποθετήσεις αποδεικνύουν ότι είμαι φιλελεύθερος. Ευχαριστώ. Σέτζο Κοφεράτη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι με την προσοχή που έχει δοθεί εδώ και τόσο καιρό στην οικονομία, τις αγορές, τις εσωτερικές σχέσεις, τις δυναμικές και τους κανόνες που θα πρέπει να τη βοηθήσουν και να τη στηρίξουν, είναι λογικό να δίνουμε τέτοια σημασία κι εμείς. Όμως, η προσοχή αυτή δεν θα πρέπει να μεταφραστεί αναγκαστικά σε νέους κανόνες και κυρίως δεν θα πρέπει να βάλουμε κατά μέρο τις πολιτικές διαστάσεις και προεκτάσεις κάποιων από τις υποθέσεις που σχολιάζουμε. Θα εξηγήσω τι εννοώ προσπαθώντας να θέσω και κάποια ερωτήματα. Τι πιστεύετε για τα προβλήματα που αφορούν την πορεία του ενίου νομίσματος της Ευρώπης. Αυτά που θίγονται με την περιθμό 4 πρόταση. Καταλαβαίνουμε την ε, ανησυχία που εδώ εκφράζεται και την καταλαβαίνουμε και τη συμμεριζόμαστε. Όμως, έχετε σκεφτεί τι θα συνέβαινε με το ενιαίο νόμισμα Εάν συγχρόνως δεν υπάρχει ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής και πραγματική επιτάχυνση ως προς την οικονομική σύγκληση, εννοώ τις φορολογικές πολιτικές που τείνουν να αποκλίνουν, αντί να συγκλίνουν. Επιπλέον, άκουσα τις παρατηρήσεις σας όταν απαντήσατε και στην πρόταση και το θέμα που έθεσε η για τους φόρους των των συναλλαγών. Προφανώς, όσο πιο μικρή είναι η περίμετρος εδώ στην οποία θα επιβάλλεται ο φόρος αυτός, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να υπάρχει διαφυγή και αρνητικές συνέπειες για την ευρύτερη αγορά. Όμως, μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό για την Ευρώπη. Κάτι που μπορεί να μην διαχειριστεί μόνη της μία χώρα, όσο μεγάλη και αν είναι, μπορεί να το διαχειριστεί καλά η Ευρώπη και να είναι χρήσιμη για την Ευρώπη. Ε, μια τέτοια κίνηση. Η Ευρώπη θα πρέπει να έχει και αυτόνομο προπολογισμό σε μια, φάση, σε μια περίοδο τέτοια μεγάλη κρίση. Φανταστείτε να καταρτίζουμε αναπτυξιακέ πολιτικέ με διαθέσιμου πόρου που είναι το σύνολο του ενεργητικού ε, κάθε ε, μεμονωμένου κράτου μέλου. Ψηφίσαμε εδώ ένα έγγραφο για στρατηγικές φιλοδοξίε έω το 2020. Χωρί αυτονομία στον προπολογισμό και χωρί πόρου, ευέλικτου μάλιστα πόρου, που να ε, συμπεριλαμβάνονται σε όσα είναι διαθέσιμα, ε, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε και πολλά χειροπιαστά αποτελέσματα. Εάν λοιπόν κάθε χώρα ξεχωριστά είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να τα καταφέρει, ίσως να μπορεί η Ευρώπη ως ε, ομάδα. Εδώ δεν θέλω μέσα από μια φιλονικία να καταλήξουμε στο να μην κάνουμε τίποτε. Διότι κάτι που ακόμη με ανησυχεί είναι η επιτάχυνση της εξέτασης κάποιων θεμάτων και η έλλειψη εξέτασης κάποιων άλλων. Το να μιλάμε για τα ευρωομόλογα, για την φορολόγηση των χρηματοδοτικών συναλλαγών, το να σκεφτόμαστε τι θα γίνει με το συνδυασμό των κρατικών χρεών. Αυτά όλα πριν από λίγους μήνες θεωρούνταν βλασφημία, αιρετικές απόψεις όχι μόνο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και ξαφνικά υπήρξε μια επιτάχυνση και αύξηση της προσοχής και της υποθυμίας όλα να τα εξετάσουμε. Χρειάζεται, λέει, υπερεθνική επαγρύπνηση. Η Επιτροπή, η Επιτροπή σας ε, συζήτησε, μάλλον η Επιτροπή μας άρχισε να συζητάμε τους προσκεκλημένους εδώ και κανείς δεν φάνηκε να διαφωνεί με την ενίσχυση της επαγρύπνησης. Όταν όμως ρωτούσαμε τον οποιονδήποτε πώς θα γινόταν η ενίσχυση αυτή, έπεφτε σιωπή. Άρα τι συμβαίνει. Πολλοί είναι πιο πρόθυμοι και προσέχουν περισσότερο και ζητούν να ε, προβλεφθούν νέα στοιχεία. Αυτές όμως οι καινοτομίες ποτέ δεν γίνονται συγκεκριμένε και χειροπιαστές. Άρα τι κινδυνεύουμε να συμβεί. Να τα κλονίσει όλα η μεγάλη αυτή κρίση, διότι οι μικρές χώρες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τις εγκαταλείψουμε, αλλά είναι σχετικά απλό να παρέμβουμε. Εάν όμως μπούμε στο σύστημα, στην ε, διαδικασία της κρίσης σε μία από τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε να αντιδράσουμε. Άρα, διερωτώ γιατί, γιατί τέτοια δυστοκία, γιατί τέτοια αδράνεια μπροστά σε ε, αυτά που πρέπει να γίνουν. Διότι φαίνεται το άλογο που πρέπει να κάνει την κούρσα τελικά να παρεκκλίνει και να πετάει και από τη σέλα από τον αναβάτη Τι θα γίνει. Θα απαντήσουμε και οι δύο, γιατί ενδεχομένως θα συμφωνούμε για κάποια ζητήματα, ενδεχομένως να αποκλείουν οι απόψεις μας για άλλα. Αν έχουμε κάποια ευθύνη, και απαντώ στον κύριο Σμιτ τώρα, για την χρηματοπιστωτική κρίση, μα ναι, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Είναι όμως αυτοί οι οποίοι μας εξήγησαν όλα αυτά τα χρόνια ότι έπρεπε να απελευθερώσουμε τις αγορές. Εγώ αισθάνομαι λιγότερο υπεύθυνο από άλλους γιατί ουδέποτε πίστευα κάτι τέτοιο. Αν καταλαβαίνόμαστε καλά. Όταν μιλάμε για απορρίθμιση, απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όταν δηλαδή καταργήσαμε πάρα πολλούς κανόνες και περιορισμούς, Υπήρχαν πάρα πολλοί τότε που λέγανε ότι ε, με λιγότερους κανόνες η αγορά μόνη της θα εξισορροπηθεί. Μα όταν καταργείται κανόνες τι περιμένετε, δεν εξισορροπούνται απόλυτα και αυτόματα οι αγορές ή μάλλον ε, εξισορροπούνται οδηγώντας σε πολύ σημαντικές κρίσεις οι οποίες όμως ε, βαρύνουν οικονομικά όχι τους χρηματοπιστωτικούς τους οργανισμούς αλλά τους ίδιους τους πολίτες. Απαντώ λοιπόν άμεσα και ειλικρινά στο ερώτημά σας. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες, είπα ότι δεν πρέπει να θεσπίζουμε κανόνες στα δημοκρατικά πολιτεύματα, κανόνες που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι σε στιγμές δυσκολιών δεν θα τους σεβαστούμε. Με άλλα λόγια θα πρέπει να θεσπίζουμε κανόνες, ναι, αλλά οι κανόνες αυτοί να είναι ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζονται και σε κάποιες ε, εξαιρετικές καταστάσεις, έτσι ώστε να μπορεί και μια κυβέρνηση να ανταποκριθεί σε μια οικονομική δυσκολία πέντι στην κοινή γνώμη και να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Κοφεράτη. Είμαι υπέρ της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το 2001 ψήφισα αντίστοιχη νομοθεσία στο δικό μου το κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο λέω απλώς είναι ότι από πολιτικής πλευράς με ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό γιατί θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παραπάνω πόρο είτε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό είτε για τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη παγκόσμιο επίπεδο, πάντως δεν θεωρώ ότι από μόνος το φόρος αυτός μπορεί να ρυθμίσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Δεν θα ρυθμιστούν αυτόματα οι χρηματοπιστωτικές αγορές μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχει ο φόρος αυτός. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν και οι αδιαφανείς συναλλαγές και τα dark pool και η φορολογική παράδοση. Παράδειση, με συγχωρείτε. Ακριβώς επειδή υπάρχουν ε, περίπου το είπαμε 80% των συναλλαγών που ξεφεύγουν από την υποχρέωση reporting, την υποχρέωση κοινοποίηση των αντολών. Δεν μπορεί δηλαδή μια τέτοια πρόταση που είναι κυρίως πολιτικής φύσης να ρυθμίσει όλη την κατάσταση. Αυτά είχα να πω εγώ κύριε Μανσέλ, έχετε τώρα το λόγο. Θα δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Ε, ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένω να διαφωνώ με τον κύριο Εμμανουέλη είναι ότι δεν υπάρχουν μόνο οι πολιτικά ηθήνοντες οι οποίοι σφάλουν, είναι και το σύνολο ουσιαστικά των ε, λαών, των πολιτών πολλοί ανάμεσά μας για πάρα πολλά χρόνια ζούσαμε με δανεικά χρήματα. Ακόμα και αν είμαστε ένα πλούσιο κράτος ή ανήκουμε σε ένα πλούσιο κράτος, δεν μπορούμε συνεχώς να ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία κερδίζουμε. Και αυτό ισχύει για πολλές χώρες, όχι μόνο για τη Γαλλία. Υπάρχει ένα έλλειμμα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι αν σαφώς το έλλειμμα είναι 75% του ΑΕΠ 60% αυτό θα μπορούσαμε να το συζητάμε όσο θέλετε. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο θα πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική εξυγίανση πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα ζουν μια κατάσταση που θα ήταν ε, μη βιώσιμη για την Ευρώπη, ας το πούμε έτσι μιλάω για πράγματα που έχουν να κάνουν με την κοινή λογική. Βλέπουμε ότι ε, πέρα από οποιασδήποτε κανόνες σταθερότητας μπορούν να υπάρχουν, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή για τις επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν σε μια χώρα για την οικονομική ανάπτυξη να στηριζόμαστε συνεχώς στον δανεισμό και στο έλλειμμα. Όσον αφορά τουλάχιστον τη Γαλλία, πιστεύω ότι θα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα δημόσια οικονομικά μας στο γρηγορότερο δυνατό και όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά τις τράπεζες, στις οποίες αναφερθήκατε και αναφερθήκατε και στο παράδειγμα Κερβιέλ, στην Επιτροπή Οικονομικών της, ε, του Γαλλικού Κοινοβουλίου πριν από δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος, σε μία ακρόαση καλέσαμε πολλούς ε, διευθυντές ε, τραπεζών για αυτό το ζήτημα ακριβώς της κερδοσκοπίας, των μηχανισμών κερδοσκοπίας κτλ. Και ένα ζήτημα το οποίο μας προκάλεσε ανησυχίες είναι ότι οι διευθυντές των τραπεζών μας είπανε και νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε πια ειλικρινά μας είπανε, κοιτάξτε, τα όσα γίνονται στην αίθουσα των σταλαγών, εγώ δεν μπορώ να τα επαληθεύσω και να τα ελέγξω. Έχω ε, υπαλλήλου που είναι μαθηματικοί, με τεράστια πείρα, οι οποίοι μου κατασκευάζουν ε, καταπληκτικά μαθηματικά μοντέλα γιατί μου επιφέρουν πάρα πολλά κέρδη και χρήματα, αλλά εγώ ίδιο ω διευθυντή τράπεζα δεν μπορώ να πω αν τα μοντέλα αυτά είναι αποτελεσματικά ή επικίνδυνα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό. και είχα πει τότε στην συναδελφό μου ότι θα ήταν πολύ καλό να καταργούσαμε κάποια από τα μέσα αυτά, όπως για παράδειγμα το high frequency trading ή το αλγοριθμικό trading, που είναι μέσα τα οποία δεν άπτονται τόσο πολύ της πραγματικότητας, είναι κυρίως κερδοσκοπικά μέσα, κερδοσκοπικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά οδηγούν στην ανάληψη συστημικών κινδύνων όσον αφορά την αγορά. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της ε, φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα να μην θέσουμε ίδια εμπόδια στον εαυτό μας. Σαφώς είναι πολύ καλό να θεσπίσουμε ένα φόρο, αλλά αν δεν το κάνουν αυτό και οι υπόλοιπε χώρες, τότε εσείς θα βρεθείτε σε μια δυσχερή θέση. Η ανταγωνιστικότητά σε παγκόσμιο επίπεδο θα θυγεί. Όσον αφορά την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το είπε και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας την προηγούμενη Δευτέρα, είπε ότι θα πρέπει εμείς να δώσουμε το παράδειγμα τροποντινά και ότι τουλάχιστον το παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν ευρωπαϊκό. Αν δεν καταφέρουμε εμείς ως Ευρωπαίοι να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για να δημιουργήσουμε το φόρο αυτό, πώς θα καταφέρουμε στη συνέχεια να πείσουμε τον υπόλοιπο κόσμο να ακολουθήσει το παράδειγμά μας. Και λέω εδώ πέρα παραθετικά ότι δεν θα πρέπει να αμφισβητούμε για εμάς τους ίδιους. Σε μια γαλλική εφημερίδα πριν από χθες ή προχθές υπήρχε μια γελιογραφία που παρουσίαζε τον κόσμο απλοποιημένο με Αμερική και Κινέζους μόνο. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να μετράμε και εμείς σε διεθνές επίπεδο. Να μπορούμε να μιλάμε ισότιμα και με την Κίνα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χάνουμε την εμπιστοσύνη που θα πρέπει λογικά να έχουμε στον εαυτό μας. Θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να μιλάμε με μία ενιαία φωνή σε διεθνές επίπεδο και θα πρέπει να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε έναν δρόμο ευρωπαϊκό τον οποίο όλοι θα ακολουθήσουμε. Ελπίζω ότι και εσείς συμφωνείτε με αυτά τα οποία λέω. Γι' αυτό κάθε φορά που μιλάμε για σύγκληση και εδώ πέρα ενδεχομένω συμφωνώ και λίγο με τον Ενρή Εμμανουελή. Αν ακολουθήσουμε μία πολιτική σύγκλησης ε, από αλληλεγγύη τότε δεν ξέρω θα πρέπει να εγγραφεί κατά αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια του γαλλικού συντάγματος. Νομίζω ότι το πέρα υπάρχει και ένα περιθώριο καλύτερης αξιολόγησης της πρότασης αυτής. Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να πετύχουμε τη σύγκληση αυτή αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το πρόβλημα όμω με τη σύγκληση αυτή είναι ότι είμαστε 27 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν ακόμα μεγάλε αποκλήσει ακόμα και στις χώρες αυτές που συμμετέχουν στην Ευρωζώνη. Μεγάλες αποκλήσεις όσον αφορά την οικονομία, τα κοινωνικά δικαιώματα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι ξεκινώντας με τη βάση αυτή είναι πολύ δύσκολο να κινηθούμε όλοι στον ίδιο δρόμο, με τον ίδιο ρυθμό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν τόσες διαφορετικές καταστάσεις από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να πετύχουμε μία ελάχιστη σύγκληση. Θα πρέπει τουλάχιστον στη Γαλλία, στη Γερμανία να καταφέρουμε στο φορολογικό τουλάχιστον τομέα να συγκλίνουμε τις προσπάθειές μας. Πριν από λίγο αναφερθήκαμε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης πιστολεπτικής ικανότητας. Δεν ξέρω είναι τόσο καλή ιδέα. Ουσιαστικά θα μπορούσαν κάποιοι εξωτερικοί επικριτές να μας πούν ότι εμείς δημιουργούμε στην Ευρώπη έναν οίκο αξιολόγησης για μας τους ίδιους, προκειμένου να μας δίνει καλούς βαθμούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν οίκοι αξιολόγησης οι οποίοι δεν έχουν κεφάλαια αναγκαστικά αγγλικά ή αμερικανικά, αλλά χρηματοδοτούνται και από χώρες όπως η Γαλλία. Το καλύτερο πιστεύω είναι να υπάρχει κατάλληλη ρυθμιστική πλαισίωση για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και είναι σημαντικό να γίνει μια πραγματική διάκριση ανάμεσα στα κράτη και τους ιδιωτικούς χρηματοπιστωτικούς φορείς στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Προσπάθησα να είμαι σύντομος στην παρέμβασή μου κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Τύρπα Τετικάινεν, παρακαλώ. Και μετά η κυρία Εντογκάλ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μελέτη που έχουμε ενώπιόν μας και έχει συνταχθεί από τους κυρίους. Ακούτε τη διερμηνία, ακούγεται η διερμηνία παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, Εδώ, σε σχέση με αυτό το θέμα, θέσατε τον δάκτυλο επί του τύπου των ύλων. Και οι προτάσεις είναι ενδιαφέρουσες επίσης. Θα ήθελα να σας ζητήσω να α, μας αποκαλύψετε περισσότερες σκέψεις για την ε, διακυβέρνηση, παγκόσμια διακυβέρνηση, τη λέσχη των 20, G20 και πώς θα μπορούσαν όλα αυτά να λειτουργήσουν. Έχετε κάποιες τέτοιες νήξεις, αναφορές στις προτάσεις σας επίσης. Παρακαλώ εσείς έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω άρρηκτα στην προηγούμενη ερώτηση και να πω κι εγώ κάτι. Δύο παρατηρήσεις θα είχα να κάνω σε σχέση με τα όσα ακούσαμε αναφέρθηκε ότι αν όλοι ομόφωνα ε, τοποθετούνται δεν είναι ομόθυμη η τοποθέτηση. Με αυτό συμφωνώ όμως θα ήθελα να αναφερθώ στους ε, εισηγητές και να πω τι γίνεται ακριβώς εδώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται για την οικονομική πολιτική. Η κύρια κατευθυντήρια γραμμή όμως είναι οι περιορισμοί που από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υιοθετούνται και ε, συστήνονται όλο και περισσότεροι περιορισμοί και περιοριστικές διατάξεις. Επαρκεί αυτή η πολιτική λιτότητας, πειθαρχίας και περιορισμών για να τελειώσει η κρίση. Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση. Η χρηματοοικονομική αγορά και οι κερδοσκοπικές αγορές συνεχίζουν να λειτουργούν και η ε, πραγματική οικονομία παρεκκλίνει από την κερδοσκοπία. Υπάρχει χάσμα μεταξύ των δύο. Δηλαδή η χρηματιστηριακή αγορά δεν συσχετίζεται πολύ με την πραγματική οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να θέσω την ερώτηση. Δεν πιστεύετε σε όποιον βαθμό ακόμα και αν συμβαίνει αυτό ότι τα στοιχεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, έχουν χαλαρωθεί. Ε, αυτό δεν βρίσκεται ως αίτιο της κρίσης. Αυτό δεν είναι το οποίο δημιούργησε και στις μεγάλες χώρες τεράστια χρέη. Τώρα τι κάνουμε. Σε πολλές περιπτώσεις ε, τα κρατικά αυτά χρέη, την κρατική υπερχρέωση δεν είμαστε σε θέση καν να τη χρηματοδοτήσουμε. Υπάρχει μεγάλος χώρος και περιθώριο για κερδοσκοπία και εμφανίζεται με διαφορετική μορφή η κερδοσκοπία στις οικονομικά αδύναμες χώρες και στις οικονομικά ισχυρές χώρες. Στα κράτη-μέλη που είναι αδύναμες χώρες αλλά είναι μέλη της Ευρωζώνης, εκεί η κερδοσκοπική επίθεση έχει αρνητικότατες επιθέσεις στο ευρώ, αρνητικότατες οι επιπτώσεις στο ευρώ και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ ότι το credit rating, rating δηλαδή ε, οίκη αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν και να είναι ανεξάρτητοι. Όμως και τα ελεγκτικά συνέδρια, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το έργο της αξιολόγησης. Και μία τελευταία ερώτηση για το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τον φόρο αυτό. Άκουσα πολλές συζητήσεις και από για αυτό το θέμα. Πολλές μελέτες δεν συντάχθηκαν έγκαιρα σε σχέση με το, το τέλος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, το, το φόρο αυτό. Πιστεύω ότι η εισαγωγή αυτού του τέλους ή του φόρου συνεπάγεται πολύ περισσότερους κινδύνους. Αλλά τίθεται εδώ το ερώτημα για ποιο αντίτιμο θα πρέπει να υποστούμε, να ανεχθούμε αυτούς τους κινδύνους. Ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα. Ερώτηση επαρκούν οι ρυθμίσεις που είναι σήμερα στη θέση τους και λειτουργούν. Και ε, τηρούνται ενδεχόμενα. Επαρκούν αυτές ώστε οι κερδοσκοπικές συναλλαγές να πάψουν και να αναχαιτιστούν στα dark pools, στις σκοτεινές αυτές δεξαμενές. Επαρκούν αυτά ή όχι. Ευχαριστώ. Εδώ δεν έχω προετοιμάσει προφανώς καμία απάντηση, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά ε, ξεφεύγουμε στη συζήτησή μας δεν πρέπει να φτάσουμε να πούμε ότι η κρίση του ευρώ προκάλεσε την ε, οικονομική κρίση. Η κρίση αρχικά είναι, δεν ήταν κρίση εμπιστοσύνης στο ευρώ. Είναι μια κρίση που αφορά τις τράπεζες, τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών και ε, δεν είναι ο ιδιωτικό τομέα σε κρίση. Μάλλον είναι ιδιωτικό τομέα σε κρίση και όχι ο, ε, οι δημόσιοι φορεί, τα κράτη που προκάλεσαν την κρίση. Αυτοί οι ιδιωτικοί φορεί είναι που κλονίστηκαν. Έπειτα οι δημόσιοι φορεί ήρθαν να ενισχύσουν, οι κρατικοί φορεί ήρθαν να ενισχύσουν του ιδιωτικού, τι τράπεζε και να ελαφρώσουν, να ελαφρώσουν το χρέο του. Όμως δεν μπορούμε να λέμε ότι το ευρώ δεν είχε καλή υγεία και βρίσκεται στην πηγή του κακού. Όχι. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα με το ευρώ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περισσότερα προβλήματα στο δολάριο. Είναι πολύ πιο χρεωμένε οι ΗΠΑ από τι ευρωπαϊκέ χώρε. Όμω, στι ΗΠΑ η κεντρική τράπεζα αγοράζει τα κρατικά ομόλογα. Άρα, ο οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν βάζουν εκείνο στο επιτόκιο για το δημόσιο χρέο, αλλά η Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, εμεί έχουμε κάνει διαφορετική επιλογή. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ευρώ, που αγορεύσαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εξαγοράζει τα δημόσια χρέη. Και στι πιο οξύε στιγμές της κρίση το έκανε αυτό, αλλά όχι ανοιχτά και μαζικά. Κατά τη δική μου την άποψη, και παραμένει προσωπική παρατήρηση, καταλαβαίνω ότι μπορεί να με τη συμμερίζεστε, αλλά για μένα δεν το έκανα με αρκετή σαφήνεια και ευθύτητα ώστε να ενθαρρύνει τι ε, χρηματοπιστωτικέ αγορέ να ορίσουν επιτόκιο. Ε, να μην ορίσουν μάλλον το επιτόκιο. Συνεχίζουν οι αγορέ να καθορίζουν το επιτόκιο. Άρα, για τα δημόσια χρέη υπάρχει συζήτηση παντού, όπω φαντάζομαι και εδώ, και το βασικό θέμα είναι ότι θα γίνει με τα ευρωμόλογα. Εγώ προσωπικός και πάλι είμαι υπέρ των ευρωομολόγων. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει σύστημα ειδικό εισόδου, ποινές, κυρώσεις, αλλά εγώ είμαι εδώ και καιρό υπέρ των ευρωομολόγων, διότι πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος το ευρώ να γίνει ένα πραγματικό διεθνές νόμισμα. Σήμερα υπάρχουν διαφορετικοί πιστωτέ παγκομίω που είμαι βέβαιο ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στι τοποθετήσει του. Και σίγουρα οι Αμερικανικέ τράπεζε θα ήθελαν πάρα πολύ να αποκτήσουν μερικά ευρώ ομόλογα για να μοιραστούν τον κίνδυνο. Λοιπόν, είναι ένας τρόπος αυτό να γίνει το ευρώ πραγματικά διεθνού βεληνικού νόμισμα. Κάτι που δεν ισχύει αναγκαστικά Τώρα, ε, λοιπόν, η οικονομία είναι ένα πολύ περίπου πράγμα. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια τη κρίση, όσοι έκαναν τοποθετήσει σε μέσα από τράπεζε, ασφαλιστικέ εταιρείε, ε, οικονομικοί φορεί, ζητούσαν κρατικά ομόλογα. Δημόσιο χρέο για να διασφαλίσουν τι τοποθετήσει του. Και είχα κάνει κάποτε μια παρατήρηση. Ευτυχώ που έχουμε έλλειμμα. Διότι δάλλως τι θα έκανε τα Πού θα βρίσκα τι ε, εγγύησει. Τα πράγματα λοιπόν ποτέ δεν είναι μαύρα ή άσπρα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βλέπει κανεί την ίδια κατάσταση. Πάντως ε, δυσκολεύομαι να υποδείξω ω υπέτειο τη κρίση το ευρώ. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό εύκολα. Είναι ένα, παραλικό, ένα παραλυπόμενο, ένα από τα θύματα μάλλον, τα παράπλευρα του ευρώ τη κρίση αυτή. Επειδή βρεθήκαμε σε αυτή τη δύσκολη θέση, επλήκει και το ευρώ τώρα για το έλλειμμα. Αυτό είναι συζήτηση πολιτικού περιεχομένου. Πρέπει να γίνει σε καμιά από τις δημοκρατικές, κάθε μια τι δημοκρατικέ μα χώρε. Χρειάζεται έλλειμμα ή όχι. Έχουμε ξεπεράσει τα μέσα διαβίωσή μα. Ναι. Μπορούμε να πούμε όμω, αγαπητέ μου Ζαν Φρανσουά, στη Γαλλία το διαφορετικό έλλειμμα των 45 έως 50 δις ευρώ ετησίως είναι το ισοδύναμο που των φορολογικών εσόδων που καταργήσαμε Γαλλοί ε, αριστεράς και δεξιάς συμπεριλαμβανομένων ε, από το 2000. Καταργήσαμε πολλούς φόρους. 45-50 δις ευρώ. Τέτοια ήταν η αξία τους. Άρα, άμα καταργείς τα φορολογικά έσοδα και δεν τα αντισταθμίσεις ή δεν μειώσεις τις δαπάνες, ε, βρίσκεσαι σε κατάσταση μη ισορροπίας. Μπορούμε να λέμε ότι ζήσαμε με περισσότερα από ό,τι είχαμε, αλλά και άσχημα τα αναδιανύμαμε αυτά που είχαμε. Ή όχι σωστά. Αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει στο επίπεδο τη κάθε χώρα. Εγώ δεν μπορώ λοιπόν εδώ να διακινδυνεύσω να κρίνω άλλου. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, να λάβω αφορμή από μια ερώτηση το κατά πόσον έχει αναχαιριστεί η κρίση. Κοιτάξτε, από άποψη οικονομική τα πράγματα βελτιώνονται συνεχώ και σταθερά. Ε, εάν δούμε τι γίνεται με την εξέλιξη των ΑΕΠ, με την βραδία ανάκαμψη τη απασχόληση, αργία αλλά σταθερή, υπάρχει μια σαφή βελτίωση. Όμω στο οικονομικό επίπεδο, στο χρηματοστοπιστικό επίπεδο δεν έχουν ε, ε, λήξει ακόμη τα προβλήματα. δείτε τις τρεις πρώτες μας προτάσεις. Επιμένουμε πάρα πολύ στην ε, μεγάλη απόκληση που υπάρχει μεταξύ της ρευστότητας, ε, έλλειψης ρευστότητας παγκοσμίω και της πραγματικότητας των ΑΕΠ σε εθνικό επίπεδο. Χοντρικά έχουμε τρεις φορές περισσότερη ρευστότητα παγκοσμίω να κυκλοφορεί παρά το σύνολο όλων των ΑΕΠ παγκοσμίω, όλων των κρατών στον κόσμο. Τη στιγμή λοιπόν θα έπρεπε κανείς να περιορίσει λίγο τη ρευστότητα για να μην υπάρχει αυτή η ροπή προς την κερδοσκοπία, εμείς θα συνεχίσουμε να την αυξάνουμε. Το είπε πριν και ο κύριος Εμμανουηλή. Ε, αυτό γιατί ακριβώ δεν υπάρχει επαρκή εμπιστοσύνη μεταξύ των τραπεζών. Δεν τολμούν οι τράπεζε να δανείσουν μια την άλλη, διότι φοβούνται ότι θα την πατήσουν, θα πάρουν τοξικά προϊόντα. Έτσι χρειαζόμαστε να τις αναχρηματοδοτούμε. Και από τη στιγμή που υπάρχει χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες, ε, ουσιαστικά ε, αυξάνουμε τη ρευστότητα. Το σύστημα είναι πολύ παράδοξο. Δηλαδή ο καθένας έχει συνέστηση ότι θα πρέπει να μειώσει την αξία της ρευστότητας που κυκλοφορεί, του ρευστού που κυκλοφορεί, αλλά συνεχώς τροφοδοτούμε την αγορά με νέο ρευστό. Διότι τα συστήματα, τα χρηματοπιστωτικά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Άρα δεν έχουμε βγει στην πραγματικότητα από την κρίση ο κύριο Εμμανουέλη και εγώ ε, έχουμε περιορισμένε εξουσίε. Δεν είναι πρωθυπουργό τη Γαλλική Δημοκρατία ο κύριο Εμμανουέλη. Μπορεί και εγώ και εκείνο να λυπούμαστε γι' αυτό, αλλά δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και να αποδείξουμε μάλλον στη θέση του κύριου Σαρκοζή. Ευχαρίστω να κάνουμε ό,τι μπορούμε με του 28 συναδέλφου μα τη Γαλλική Βουλή. Θα ετοιμάσουμε δηλαδή την έκθεση για την οικονομική κερδοσκοπία και ποιε ήταν οι αρνητικέ τη συνέπειε και ποιε θα είναι και στο μέλλον. Για την ζωή τη πραγματική οικονομία, τη ζωή των ε, πολιτών μα ως οικονομικών φορέων. Μόνο τέτοιε απαντήσει μπορούμε να σα δώσουμε τώρα. Αυτέ οι ερωτήσει που θέτετε είναι πολύ συμπαθητικέ, όμω για την διεθνή διακυβέρνηση υπάρχουν απαντήσει ω πολιτικοί ευθύνοντε. Κάτι μπορούμε να πούμε, αλλά δεν μπορούμε να σα δώσουμε και παγκόσμιου ελληνικού απαντήσει. Πάντω, ειλικρινώ νομίζω ότι αν εδώ καταφέρναμε ένα μέρος των προτάσεων τη Επιτροπής σα, κύριε Πρόεδρε, με του συναδέλφου σα, ένα μέρο των προτάσεων αυτών που εμεί κάναμε στο επίπεδο τη Εξεταστική μα Επιτροπή, εάν ένα μέρο όλων αυτών εφαρμόζονταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνέ, οπωσδήποτε θα είχαμε κάνει ένα άλμα, ένα τεράστιο βήμα προ την παγκόσμια διακυβέρνηση για την οικονομική και χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως επιτρέψτε μου και εμένα στο τέλο να κάνω κι εγώ ένα-δύο σχόλια και να αναφερθώ και να διατυπώσω δύο-τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, το πεδίο εξέτασης της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ήταν ευρύτερο από το δικό σας. Δεν ασχοληθήκαμε μόνο με θέματα της κερδοσκοπίας και της οικονομικής κρίσης στο στενότερο πλαίσιο, αλλά θέλαμε ουσιαστικά όσο γινόταν, όσο περισσότερο σε ευρύτερο πλαίσιο γινόταν να ξεπεράσουμε αυτά τα πλαίσια για τα οικονομικά αίτια. Όσον αφορά τα αίτια, μόνο εν μέρη, κύριε Εμμανουελή, συμφωνώ μαζί σας. Φυσικά όλα αυτά άσκησαν, είχαν την επιρροή τους στον ε, τομέα των ακινήτων στην ε, Αμερική, στη ΣΥΠΑ και τα subprimes. Αλλά είναι και πολιτική η εμπλοκή. Η στοχοθέτηση της Αμερικανικής κυβέρνησης, κάθε πολίτης να έχει το δικό του διαμέρισμα με δάνεια, με πιστώσεις, μάλιστα και η δυσανάλογη, δυσανάλογα χαλαρή πολιτική για χορήγηση δανείων με υποθήκες, υποθήκες των ακινήτων ε, είναι όλα αυτά που οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Ακαθώς επίσης και οι εποπτικές αρχές. Η αποτυχία τους στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη είναι εξόφθαλμη. Πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα. Και τα λανθασμένα κίνητρα όσον αφορά ε, το σύστημα που υιοθετήθηκε και η κερδοσκοπία, αλλά όχι μόνο η κερδοσκοπία, κύρια και μόνο η κερδοσκοπία, έχουν συνταχθεί και διαφορετικές μελέτες για τις επιπτώσεις της κερδοσκοπίας, ακριβώς όσον αφορά το, την κρατική υπερχρέωση, το κρατικό χρέος της Ελλάδας. Και τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά, μας εξέπληξαν, διότι έλεγαν αυτά τα αποτελέσματα ότι ουσιαστικά η κερδοσκοπία δεν είχε τέτοιες μεγάλες επιπτώσεις, ήταν ελάχιστη η επίπτωσή της. Και δεύτερον, δεν πρέπει, δεν επιτρέπεται να ξεχνάμε ότι το ευρώ σίγουρα δεν είναι το αίτιο της κρίσης. Σίγουρα συμφωνούμε απόλυτα επ' αυτού. Α, συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι κάθε, κάποια μέλη της Ευρωζώνης για πολλά χρόνια για μεγάλο χρονικό διάστημα ακολούθησαν μια ανεύθυνη πολιτική που υιοθέτησαν. Όταν ακούμε ότι στην Ελλάδα οι μισθοί σε 10 χρόνια αυξήθηκαν 54%. Κάθε χρόνο αυξανόντουσαν 5,4%. Πολύ περισσότερο αυξανόντουσαν από τη αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη ότι είχε προβλήματα η παραγωγικότητα και το ρυθμός ανάπτυξης. Ε, αυτό δημιούργησε προβλήματα. Αυτό δεν έχει σχέση με το ευρώ θεωρώ ούτε έχει σχέση με κάποια κερδοσκοπία, αλλά είναι λανθασμένη πολιτική που ακολουθήθηκε. Εντάξει, παρέμβαση χωρί μικρόφωνο δεν ακούγεται. Φυσικά λέει ο πρόεδρο και συνεχίζει. Αλλά είναι γεγονό ότι οι κοινωνικοί εταίροι στην Ελλάδα έκαναν κάποιες συμφωνίες που από οικονομικής πλευρά έκαναν μια πολιτική που δεν μπορούσε να ε, είναι βιώσιμη με ε, τα στοιχεία που έχουμε. Πολύ σωστό αυτό, όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε τώρα ότι η γαλλική τράπεζα και στην ε, Γερμανία το ίδιο συμβαίνει. Οι Γάλλοι εμπλέκονται ιδιαίτερα για τις, ε, την αγορά ε, ομολόγων από την Ελλάδα, από την Πορτογαλία και άλλα. Αν δεν επιστραφούν αυτά τα κονδύλια και αν δεν υπάρχουν προοπτικές για κάτι τέτοιο, έστω και με κούρεμα, δηλαδή με, ε, το να κουρέψουν, να, μειωθούν, ε, η, να μειωθεί η υπερχρέωση, τότε δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Έρχομαι στην ερώτησή μου τώρα. Γνωρίζουμε ότι οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, απέχουν όλο και περισσότερο από την Ευρώπη δεν είναι πια φιλοευρωπαίοι όπως ήταν κάποτε στο παρελθόν. Ούτε είναι πισμένοι πια ότι η Ευρώπη είναι το μέλλον τους. Δυσπιστούν πολύ και αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Διότι αυτό είναι η βάση ξαφνικά πάλι να καταλήξουμε σε εθνικοποιημένες πολιτικές, στην επανεθνικοποιημένη στροφή ε, εθνικών πολιτικών και αυτό είναι επικίνδυνο. Ερωτώ λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε κύριοι ώστε πραγματικά να μπορέσουν οι πολίτες να ταυτιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να βελτιωθεί η κατάσταση, να έρθουν πιο κοντά προς την Ευρώπη οι πολίτες. Δεύτερον, γνωρίζουμε όλοι ότι στο μέλλον χρειάζεται ανάπτυξη. Χωρίς ανάπτυξη, μόνο με ρυθμίσεις και περιορισμούς δεν θα κάνουμε τίποτα. Χρειαζόμαστε φιλική Κύπρος στις επενδύσεις ε, πολιτική και ένα κλίμα θετικό για να αντιμετωπιστούν τα χρέη. Χωρίς ανάπτυξη δεν θα έχουμε τα κονδύλια για να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Χωρίς επενδύσεις για το μέλλον θα είμαστε πραγματικά, ε, ας το πω έτσι, δεν θα είμαστε στην ομάδα των τριών ή τεσσάρων μεταξύ των ΙΠΑ, τη ε, της Βραζιλίας, της Κίνας και των άλλων μεγάλων, αλλά θα είμαστε πλέον στη δεύτερη κατηγορία. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε τουλάχιστον να διασφαλίσουμε αυτή την πτυχή για το μέλλον. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα απαντήσουμε ξεχωριστά όμως αυτή τη φορά νομίζω. Ενδεχομένως κάπου να συγκλίνουν οι απόψεις μας, κάπου να συναντηθούμε στο δρόμο, αλλά θα απαντήσω εγώ καταρχάς για την κρίση. Πρόκειται για μια χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία οφείλεται σε μια δανειοδοτική πολιτική που ακολουθήθηκε είτε ανεύθυνη όπως με τα subprimes είτε ιδιαίτερα έντονη αν θέλετε, είναι μια πολιτική την οποία εμείς οι ίδιοι ενθαρρύναμε. Και δεν φταίει αναγκαστικά η Αμερικανική, η Γαλλική, η Γερμανική κυβέρνηση. Δεν είπαν οι κυβερνήσει ότι πρέπει να δώσετε περισσότερα δάνεια. Αυτό το οποίο συμβαίνει όμω στην πράξη, και τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, ενδεχομένω κάποιοι διαφωνούν μαζί μου, όταν όμως βλέπουμε ότι η αναδιανομή των κερδών μεταξύ μισθωτών και μετόχων δεν γίνανε, δεν έγινε με το σωστό τρόπο, βλέπουμε ότι οδηγηθήκαμε ουσιαστικά σε μία έντονη δανειοδότηση η οποία ήρθε να αντισταθμίσει την ε, κακή αναδιανομή του πλούτου, του κεφαλαίου. Σαφώς μπορεί άλλοι πολιτικοί να έχουν διαφορετική τοποθέτηση. Δεν φταίει λοιπόν το ευρώ. Για το ευρώ βέβαια είχαμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές καταστάσεις. Χώρες οι οποίες μπήκαν στην ευρωζώνη μια δεδομένη στιγμή και βρισκόντουσαν σε διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και που στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς γνώρισαν ένα έντονο φορολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ, ναι, είναι χώρες οι οποίες υπέφεραν. Οι χώρες όμως αυτές γνώρισαν τον ντάμπινγκ αυτό ακριβώς επειδή η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έγινε με τον ίδιο ρυθμό που είχε γίνει στο παρελθόν. Η διεύρυνση που είχε γίνει με την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις πρώτες χώρες ήταν μια διαδικασία πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο όρημη. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, με τη δεύτερη διεύρυνση δεν είχαμε τα απαραίτητα χρήματα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε την απαραίτητη αναδιανομή κεφαλαίων. Είπαμε λοιπόν στις χώρες αυτές, κοιτάξτε δεν έχουμε χρήματα να σας δώσουμε, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας και βέβαια κατέληξαν σε κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ. Σαφώς λοιπόν όλοι φέρουμε ευθύνες για αυτά τα οποία συνέβησαν στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Και δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί κάποια μέρα το ευρώ, ότι θα καταρρεύσει. Διαβάζουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και κάποιες ανοσίες αν θέλετε για το ζήτημα αυτό τελευταία. συνεχίζω και έχω εμπιστοσύνη στην ε, ικανότητα των ευρωπαϊκών κρατών να τα βγάλουν πέρα. Και να έρθω κατευθείαν στο ερώτημα του Πρόεδρου, του πρόεδρου σας. Η οικονομική ανάπτυξη, σαφώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε οποιοδήποτε δάνειο αν δεν υπάρχει οικονομική ανάπτυξη. Όσο και να μειώσουμε το χρέος και το έλλειμμα, αν δεν καταφέρουμε να κτίσουμε την οικονομική μας ανάπτυξη, δεν πρόκειται να τα βγάλουμε πέρα. Ή θα γίνει, αν θέλετε, πραγματικά μία... Θα έχουμε μία θα έχουμε πολύ δυσάρεστε οικονομικέ εξελίξει. Μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για πραξικόπημα εντό αγωγικών, πολιτική φύσεω, αν τυχόν δεν καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα έχουμε παρεκκλήσει πάρα πολύ έντονε και ανυπόφορε πολλέ φορέ για του πολίτε. Επομένω, πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια κατάσταση οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει κάθε φορά που υπάρχει ένα κοινό σχέδιο να σταματάμε πλέον να τρογόμαστε μεταξύ μας για τη χρηματοδότηση. Βλέπουμε ότι όλα τα ευρωπαϊκά σημαντικά σχέδια αυτή τη στιγμή δεν προχωρούν ακριβώς επειδή δεν καταφέρνουν μεταξύ μας να εγκρίνουμε τη χρηματοδότησή τους. Πρέπει λοιπόν μαζί να καταφέρουμε να κάνουμε διάφορα πράγματα, πρέπει μαζί να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, εφόσον λοιπόν συμφωνούμε για ποιο λόγο δεν χρηματοδοτούμε τα απαραίτητα σχέδια. Όταν φτάνουμε στο κεφάλαιο αυτό τη χρηματοδότηση ξαφνικά δεν βρίσκουμε του απαραίτητους πόρου για να χρηματοδοτήσουμε τα, τα σχέδια αυτά. Και αυτό πραγματικά είναι ε, απαράδεκτο, είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Και δεν θα πρέπει να δημιουργούμε όλο και περισσότερο μία Ευρώπη που να παρουσιάζει ένα τεράστιο, ένα τεράστιο κενό. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι διαπραγματευόμαστε με την Κορέα, 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Ευρώπη είναι 500 εκατομμύρια πολίτες. Και αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέτουμε εμείς κανέναν όρο αντισταθμιστικό, δεχόμαστε την αχαλήνοτη εισαγωγή προϊόντων αυτοκινήτων, συγκεκριμένα από την Κορέα. Μα γιατί το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ήδη αρκετά νοσηρή η οικονομική μας κατάσταση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Δείτε τι γίνεται για παράδειγμα με τον Καναδά και στις σχέσεις που έχει ο Καναδάς και με το Μεξικό ή δείτε τις σχέσεις Μεξικού Ηνωμένων Πολιτειών. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα ήθελα να πιστοδρομήσουμε, αλλά με λυπεί το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να υπεραμεινθεί του βιομηχανικού της τομέα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, και δεν αναφέρομαι μόνο στο γαλλικό, στη, στη Γαλλία, αναφέρομαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν βλέπουμε ότι περισσότερε περισσότερες ευρωπαϊκές βρίσκονται σε δύσκολη, δεινή οικονομική για ποιο λόγο ακολουθούμε εμείς αυτή την πολιτική. Για ποιο λόγο βγαίνουμε και λέμε προς όλο τον κόσμο προς τα έξω ότι σας προσφέρουμε εμείς την ελεύθερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, σαν να θέλουμε πάση θυσία να ικανοποιήσουμε τις τρίτες χώρες. Σαφώς μπορεί ορισμένοι να εποφελούνται από την πολιτική αυτή, αλλά αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να υποφέρει το σύνολο του βιομηχανικού τομέα. Όταν λέτε λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο, συμφωνώ ναι, πρέπει να έχουμε όμως πρώτα κοινά σχέδια, να χρηματοδοτήσουμε τα κοινά αυτά σχέδια, να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της καινοτομίας και να σταματήσουμε επιτέλους να είμαστε μία ήπειρος που έρχονται όλοι οι επιχειρηματίες για να δραστηριοποιηθούν οικονομικά εκτός από εμά. Ευχαριστώ. Σε αυτό ακριβώς καταλήγουμε ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποια κοινά σχέδια και να τα χρηματοδοτήσουμε και ότι θα πρέπει ακριβώς να εκδώσουμε κοινά ομόλογα ευρωπαϊκά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε ευχαριστώ, Περβάνς, που μου δίνεις το λόγο για λίγα δευτερόλεπτα. Όπως είπε ο Άρη, εδώ ίσως να ξανασυμφωνήσουμε. Πρόεδρε, σε αυτό που είπατε και εσείς ο ίδιος, θα πρέπει να έρθω και εγώ να προσθέσω τη δική μου τη φωνή για το ερωτηματολόγιο που μας απευθύνατε μας παρομοιάζεται λίγο με χωροφύλακες που θέλουν να νουθετήσουν, να ρυθμίσουν. Όχι, δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη και δική μας πατρότητα. Θεωρούμε ότι είναι το μόνο μέσο που μπορεί να επιτρέψει στις πραγματικές οικονομίες να λειτουργήσουν πιο εύρυθμα ε, προς όφελος των συμπολιτών μας. Όμως το πραγματικό θέμα είναι εκεί που και εσείς το θέσατε και το έκανε αυτό και ο κύριος Εμμανουελή. Δηλαδή η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει ε, το ποσοστά ανάπτυξης που δεν είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τους βασικούς μας ανταγωνιστές παγκοσμίω. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε όλοι για να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή, όχι για να φτάσουμε την Κίνα, έχει άλλα ποσοστά ανάπτυξη, αλλά να έχουμε τέτοια επίπεδα ανάπτυξη που να μα ελαφρώσουν από το χρέο, αλλά επιτρέψουν και στου πολίτε μα, στου συμπολίτε μα να ζουν καλύτερα. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Όλα τα ερωτήματα σα είναι εύστοχα. Μπορούμε να διερωτώμαστε για τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει μια λύση. Ίσως υπάρχει ένα καλό χρέος σε σχέση με το κακό αυτό χρέος που προηγουμένως σχολιάζαμε, ίσως αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε και να αυξήσουμε την παραγωγή μας και έτσι οι Ευρωπαίοι συμπολίτε, όπου και αν κατοικούν στην επικράτεια των 27, να μπορούν να βελτιώσουν τη διαβίωσή τους όσο το δυνατόν συντομότερα, σε καθημερινό επίπεδο. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση. Σε ευχαριστώ, Περβάνς, που μου άφησες αυτή την ευκαιρία να παρέμβω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Για την ε, μία και μόνη οδό που αναφέρατε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά ή αν είναι πολύ νωρίς. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτό που κάνουμε είναι και λίγο και καθυστερημένα έχουμε ξεκινήσει. Κάθε φορά που κάτι κάνουμε. Τώρα, οργανώνοντας το G20, και ενώ έχουμε τον παλάκι στα χέρια μας. Το να μην έχουμε νέα φωνή ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόβλημα. Δεν είπατε ότι διαφωνείτε προς αυτό το θέμα, αλλά από τα λόγια σας αυτό φάνηκε. Ο κύριος Εμμανουελή μας είπε όχι ενιαία φωνή για το ευρώ χωρίς δημοκρατικό έλεγχο για να βασιστούμε, ενώ ο κύριος Μασέλ είπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να έχουμε κύρος απέναντι στο G2. Εδώ φαίνεται να υπάρχει ένας βηματισμός λίγο περίεργος που δεν ξέρω αν μας οδηγεί σε πρόοδο σε χώριση για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εγώ αυτό που θέλω να σκεφτούμε είναι ότι σήμερα έχουμε φτάσει πια στην κρίσιμη μέρα. Και αυτό ξεπερνά λίγο το πλαίσιο τη συζήτησή μα για την κερδοσκοπία. Βλέπουμε πολύ καλά ότι αυτό που φτιάχνουμε, αυτό που μα στορεύουμε, δηλαδή τη διάσωση τη Ευρωζώνη, δεν ε, δίνει λύση στο ερώτημα, στο πρόβλημα, στη διαπίστωση ότι υπάρχει δηλειτουργία στην Ευρωζώνη. Το πρόβλημά μου λοιπόν, και θα επαναλάβω ή θα αφορμή από κάτι που υπόθηκε προηγουμένω, εκτό αν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί, για την δημοκρατική λειτουργία και το τι κάνουμε σήμερα. Δεν πρέπει εδώ να βρούμε κάποιε απαντήσει. Διότι η Ευρωζώνη προφανώ δεν είναι υπεύθυνη για την κρίση, αλλά είναι θύμα τη. Αυτό κανεί δεν το αρνείται. Είναι θύμα τη κρίση και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο. Δηλαδή, αυτά που αρχικά τη στήριξαν, το Σύμφωνο Σταθερότητα, ότι δεν υπάρχει στήριξη, σύγκληση στι οικονομικέ πολιτικέ, όλα αυτά την αναγκάζουν να πληρώσει ένα βαρό, βαρύ τίμημα λόγω της κρίσης. Αν όλα αυτά λοιπόν δεν οφείλονται στις ε, σχέσεις που έχει δημιουργήσει η κρίση και στην ανάγκη αντίδραση στην κρίση θα έχουμε χάσει μια ευκαιρία. Το να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, κάτι που επιδοματικά το κάναμε, με ιδιαίτερη έμφαση μάλλον το κάναμε στην Επιτροπή της Επιτροπής μας, ε, να πω ότι το κάναμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος ομοσπονδιακός φεντεραλιστικός στην έκθεση προκειμένου να μην ε, έχουμε και παρεμβολές θεσμικές. Με τους ε, συναδέλφους της ομάδας των σοσιαλιστών μου είπαν ότι σε καθένα από τα ομοσπονδιακά κράτη η Washington ε, είναι απεχθής Άρα δεν ήταν εκεί το θέμα, ούτε θέλαμε να θίξουμε τέσσερι ευαισθησίε. Πολλά μπορούμε να επικρίνουμε στις ΗΠΑ, νομίζω. Αλλά τον πρόεδρο τον εκλέγουν όλοι. Χωρί άμεσο έλεγχο, βεβαίω και το καθεξή. Α αναρωτηθούμε λοιπόν. Το να μην θέσουμε αυτό το ερώτημα σημαίνει ότι βάζουμε τρικλοποδιά μόνοι μα στον εαυτό μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχει κοινέ αρμοδιότητε, δεν τι ασκεί παρά μόνο για τη διοργάνωση της εσωτερικής αγοράς, αλλά χωρίς στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής. Και εάν δεν κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα που τόσο πολύ γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε, το μόνο που κάνουμε είναι να λέμε συνεχώ χρειαζόμαστε και άλλο συντονισμό. Εγώ από τότε που άρχισα να ασχολούμαι με το ευρώ και επειδή έχω ασχοληθεί από το Μάστεχτ και μετά είναι αρκετά τα χρόνια πλέον, συνηγορούσα υπέρ τη περισσότερη του περισσότερου συντονισμού των ε, οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Άρχισα να κουράζομαι, μπούχτησα με αυτή τη στρατηγική. Ε, αναλαμβάνω την ευθύνη. Αυτό που και ο συνάδελφος ε, είπε ότι δεν θα λειτουργήσει, ότι δεν αρκεί ο συντονισμός, ότι είναι παρεμβατικό ο συντονισμό για τι μικρέ οικονομίε των αδύναμων χωρών από ότι για τι ομοσπονδιακέ χώρε που είναι μεγαλύτερε και εκεί δεν είναι τόσο αποτελεσματικό ο συντονισμό. Με συγχωρείτε που τόσο πολύ διευρύνω το πεδίο τη συζήτησή μα, αλλά νομίζω ότι υπό το φω τη ε, προοπτική να φτάσουμε στο G20, τη προοπτική να πορευτούμε σε στρατηγικέ ε, μακροπρόθεσμων επενδύσεων ε, για τα θέματα αυτά, Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Και τώρα για τους τεχνικούς όρους που είναι πιο πεζοί αλλά έχουν τη σημασία τους. Με εξέπλησε η πρότασή σας υπαριθμών 24, διότι τώρα είχα την εντύπωση ότι στη Γαλλία αυτό ήταν ταμπού. Καταλαβαίνω όμως ε, ότι ε, ο διαχωρισμός των τραπεζών χρεογράφων και των τραπεζών ε, των επιχειρήσεων είναι κάτι που το καταφέρατε ακόμη και αν έρχεστε από διαφορετικέ πολιτικέ παρατάξει με την ένωσή σα. Λοιπόν, για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, εγώ ε, συμπαρατάσσομαι με αυτού που λένε ότι μπορεί και χρήσιμο να είναι ένα τέτοιο φόρο για να έχουμε νέε πηγέ εσόδων, για να τροφοδοτήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, για τι μακροπρόθεσμε επενδύσει και άλλα. Ε, δεν θα συγκρίνω τώρα όλα αυτά μεταξύ του, αλλά και για την ρύθμιση. Νομίζω ότι η φορολόγηση των χρηματοδοτικών ε, συναλλαγών πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως ένα ισοδύναμο του ΦΠΑ για τα εμπορεύματα. Δηλαδή, εάν επιβληθεί στον καθέναν από τους φορείς, θα δίνει επαρκή διαφάνεια στις συναλλαγές που διενεργούνται και αν θέλετε να καταπολεμήσετε το ε, high frequency trading, ε, μην μου πείτε ότι δεν είναι αυτός ο αποτελεσματικός τρόπος, ο καλύτερος τρόπος να σκοτώσουμε το high frequency trading είναι να υπερβάλλουμε ε, στους υπολογιστές που κυκλοφορούν στην αγορά να έχουν και ένα μικρό που ε, θα παρακολουθεί. Ε, ο κάθε κερβιέλ και ο καθένας των αυτών δεν θα μπορούν να παρακάμψουν ένα τέτοιο σύστημα. Θα μπαίνουμε λοιπόν στις αγορές αυτές και το μόνο που θα έχουμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε το μικροτσίπ λειτουργεί σωστά. Αυτές είναι οι δικέ μου πρώτες σκέψεις. Αλλά αν εμεί ω νομοθέτε δυσκολευόμαστε και πνιγόμαστε με τις τόσες νέες τεχνολογίες που μας προσφέρονται και αρνούμαστε αυτή την πρόκληση. Να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη, ενώ έχουμε τόσα αριθμιστικά μέσα στη διάθεσή μας. Ε, κρίμα θα είναι. Και τελευταία παρατήρηση μάλλον, όταν λέτε ότι υπάρχει κόποση. Υπάρχει κόποση από την ε, Έλλειψη υλοποίηση. Να σα θυμίσω τι έγινε την περασμένη εβδομάδα όμω. Με τι ε, εποπτικέ αρχέ που με τόση δυσκολία καταλήξαμε να δημιουργήσουμε υπό τη δίκαιη και σωστή όθηση που μα έδεσε ο κ. Λαροζιέρη. Πολεμήσαμε για να έχουν οι αρχές αυτές πραγματικές εξουσίες. Και σήμερα τι βλέπουμε. Τα μεγάλα κράτη-μέλη δεν θέλουν να παίξουν αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Δεν διόρισαν πρόσωπα για να διευθύνουν τις αρχές αυτές. Και θα ξεκινήσουμε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή ζηλόφθονα κρατάει τις εξουσίες της και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη, Κανεί, λοιπόν δεν σκέφτεται τι αρχικά ξεκινήσαμε να κάνουμε. Όταν θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια εποπτική αρχή ευρωπαϊκή με συγκεκριμένε αρμοδιότητε σε ευρωπαϊκή εμβέλεια, δημιουργήσαμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δέκα χρόνια πριν υπήρχε το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών ε, Μελετών και αναγνωρίζεται πλέον με το κύρος της η τράπεζα αυτή σήμερα, ενώ τώρα θέλουμε εποπτικές αρχές ε, για τις χρηματοπιστικές αξίε και τα μεσητικά, ε, έχουμε πάλι μια εμπειρία δεκαετίας πίσω μας στην ανάλογη επιτροπή και πλέον υποβαθμίζουμε οι ίδιοι τα μέσα που διαθέτουμε και ω προ τα κονδύλια και τον προπολογισμό και το προσωπικό των αρχών αυτών. Να λοιπόν, κάτι που θα πρέπει να σας ε, χτυπήσει συναγερμό ε, ως Επιτροπή, αρμόδια, ως Επιτροπή Αρμόδια για τα θέματα της ε, κερδοσκοπίας. Ε, ευρωπαϊκές αρχές είχαμε τέτοιες ευκαιρίε και νομίζω ότι τις χάνουμε και εξαιτία των κρατών μελών και τη Επιτροπή του βάζω και του δύο στο ίδιο τσουβάλι γιατί έχουν κάνει τα ίδια. Εμεί πολεμήσαμε ιδιαίτερα ώστε οι τρει αρχέ αυτέ για τι τράπεζε, τι ασφάλειε και τι κινητέ αξίε να έχουν πραγματικέ εξουσίε. Αλλά απεχθάνεται Τη σκέψη δημιουργία τέτοιων αρχών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ω τώρα εκείνη μπορούσε να κάνει τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε μόνη τη και ούτω καθεξή. Εμεί αγωνιστήκαμε, δώσαμε μάχη για να έχουν και αυτόνομη, ανεξάρτητη ρυθμιστική λειτουργία οι αρχέ αυτέ. Τα κατημέλη δεν πρικοδότησαν με τον απαραίτητο προπολογισμό τη αρχή αυτέ, ώστε να μπορούν να στρατολογήσουν τα άτομα αυτά που θα είναι σε θέση να σκεφτούν και να βρουν τον καρδιέλ. Άρα για να υπάρχει αρχή ευρωπαϊκή με ανάλογες εξουσίες όπως η γαλλική εποπτική αρχή, θα έπρεπε να έχει γίνει κάτι ανάλογο. Όμω, ποιοι διορίστηκαν. Θα σα τα πω γαλλικά για να καταλάβετε καλά. Αυτό που διορίστηκε υπεύθυνο τη ΣΜΑ, τη αρχή που είναι υπεύθυνη για τι κινητέ αξίε, είναι κάποιο που ο κ. Ζουγέ δεν γνώριζε την παραμονή τη διορισμού του. Την αρχή δηλαδή του τομέα του δεν ξέρει ποιο την διευθύνει. Ε. Θέλετε να προσθέσετε τίποτα άλλο. Όχι. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν της συναδρίασής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε.